τα προβλήματα του να καταμετράμε. Και επίσης... Ποιος δεν έχει φέρει την κάρτα του, την κάρτα ψηφοφορίας. Εντάξει, εντάξει, θα το έχουμε υπόψη μας. Άλλος. Δεν είναι καλά παιδιά οι βουλευτές μου φαίνεται σήμερα, λέει η πρόεδρος. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσουμε με ηλεκτρονική ψηφοφορία και θα καταγράψουμε και αυτούς που δεν είχαν την κάρτα τους μαζί τους. Και ελπίζω θα λειτουργήσει γιατί αλλιώς με αυτή την κυκλική αίθουσα είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε σε ποια πολιτική ομάδα ανήκει ο καθένας σας. Λοιπόν, ηλεκτρονικά. Έχουμε τρία άτομα τα οποία δεν έχουν την κάρτα τους. Ο κύριος αυτός από το ΕΛΚΑ, η κυρία Ανδρές Μπαρέα και ο κύριος Χάντο. Όταν την έχετε την κάρτα σας, όταν σας τη φέρουν, πέστε μας για να μην μπερδευτούμε. Ξεκινάμε λοιπόν. Έχουμε τρεις ψηφοφορίες που είναι <clears throat> κατευθυντήριο χαρακτήρα. Καταρχήν Έχουμε τη μεγάλη χαρά να πούμε ότι για πρώτη φορά λειτουργούμε σε επίπεδο συναπόφασης με την συνθήκη της Λισαβόνας η οποία ετέθη σε εφαρμογή. Είμαστε για πρώτη φορά λοιπόν μια συνομοθετική επιτροπή. Και οι, τρίτες, οι ψηφοφορίες, οι τρεις είναι απλώς ψηφοφορίες για να δώσουμε εντολή διαπραγματευτική στους εισηγητές μας που πρέπει να διαπραγματευτούν με το Συμβούλιο. Είναι απαραίτητο να υπάρξει λοιπόν αυτή η ψηφοφορία για την ανάγνωση, την πρώτη ανάγνωση των τριών αυτών εκθέσεων. Όπως ξέρετε, στις διαπραγματεύσεις πέραν του εισηγητού θα είναι παρόντες και οι σκιώδεις εισηγητές, δεν πρόκειται να τους αναφέρω. Ξέρετε ποιοι είναι οι σκιώδεις εισηγητές για αυτές τις τρεις εκθέσεις και μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν ήδη στην αρχή της ψηφοφορίας. Ξεκινάμε με τη δική μου έκθεση σε σχέση με την ε, πολυμερή συνεργασία στο Βόρειο Ατλαντικό. Έχουμε τις τροπολογίες της δικιάς μου και τις τροπολογίες του κυρίου Φερέιρα. Εγώ είμαι υπέρ της τροπολογίας. Ποια είναι αυτή η τροπολογία τώρα να θυμάμαι. Τρία. Για την 11 είμαι κατά. Και για την τελευταία τροπολογία είμαι κατά. Όχι γιατί δεν θέλω να αναφέρεται ο κανονισμός της, ε, της ε, ακανόνιστης και παράνομης αλληλείας, αλλά διότι δεν έχει νόημα να επαναλαμβάνουμε συνέχεια τον κανονισμό αυτό. Ξεκινά λοιπόν με την τροπολογία 1. Ψήφι υπέρ. Δύο Ψήφι υπέρ. Eh, eh, ψηφίζουμε την έκθεση Φράγα και ξεκινάμε με την τροπολογία υπαριθμών 1 και θέτω σε ψηφοφορία την τροπολογία υπαριθμών 1. Άρχεται η ψηφοφορία και όσοι δεν έχουν κάρτα <clears throat> να μας πούν πώς ψηφίζουν. Κύριε Φάλλον παρόν. Έχω, έχω, έχω, έχω τώρα κάρτα. Κύριος Χάνο θα μας λέει ποια είναι η θέση του. Λοιπόν, πέρας ψηφοφορίας. 12 ψήφισαν, 13 <clears throat> με, τις, ε, με την κάρτα που λείπει. 13-0 εγκρίνεται λοιπόν η τροπολογία αυτή. Η τροπολογία 2. άρχιτη ψηφοφορία. Δεκαπέντε ψήφισαν και 15 υπέρ. <clears throat> Τροπολογία 10. Φερέιρα. Άρχεται ψηφοφορία. Λήξεις. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία και πάλι σας λέω. Δεν ξέρω με ποιο κατάλογο ψηφοφορία ψηφίζετε εσεί. Εγώ έχω τον κανονικό κατάλογο. Είναι πολύ δύσκολο να καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα που έχετε. Τροπολογία 10 σα υπάρχει την ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. 16 ψήφισαν, 12 υπέρ, 2 κατά και 2 αποχές. Εγκρίνεται τροπολογία. Συνεχίζουμε. Ψηφοφορία της τροπολογίας υπαριθμών 3. Άρχεται. Σε cierra la votación. Πέρας. 16 ψήφισαν, 15 υπέρ, κανείς κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Άρχεται ψηφοφορία. Σε 16 ψήφισαν, 16 υπέρ. Τροπολογία 11. Φερρέιρα. Άρχεται την ψηφοφορία. Πέρασε. 17 ψήφισαν και 17 κατά απορρίπτεται η τροπολογία. Τροπολογία 5. Πέρας. Δεκαεπτά ψήφισαν, 7 υπέρ, και τέσσερις ε, απόχες εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Πέρας ψηφοφορίας. 10 εξψήφισαν, 13 πέρα, 3 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας. 17 ψήφισαν, 17 υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Πέρας. 17 ψήφισαν, 16 υπέρ, μια αποχή εγκρίνεται, η 8. Η τροπολογία 12 τώρα του κυρίου Φερέιρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. 17 ψήφισαν 5 υπέρ και 12 κατά. Απορρίπτεται η τροπολογία. Τροπολογία 9. Πέρας. 17 ψήφισαν, 17 υπέρ η τροπολογία αυτή. Και έρχομαι τώρα στην τροπολογία υπαριθμών 1, η προφορική τροπολογία. <clears throat> Είναι για να προσαρμόσουμε τα άρθρα αυτά της έκθεσης στη νέα διαδικασία επιτροπολογίας που προβλέπεται από την Συνδίκη της Λισαβόνας. Έχετε το κείμενο της τροπολογίας, αλλά σας εξηγώ ποιος είναι ο στόχος της. Θέτω σε ψηφοφορία λοιπόν την τροπολογία 1. Προφορική. Ψήφι υπέρ. Άρχια την ψηφοφορία. Μάλλον πέρα ψηφοφορία 17 ψήφι, 17 υπέρ. Ενεκρίθη λοιπόν ομόφωνα αυτή η τροπολογία. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους. Τελείωσε λοιπόν αυτή η ψηφοφορία κατεύθυνση. Περνάμε στην επόμενη έκθεση που είναι η έκθεση της κυρίας Μπιλμπάου Μπαραντίκα για, το, για τον Γάβρο. Έχει το λόγο η κυρία Μπιλμπόα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στον κατάλογο ψηφοφορίας που έχουμε διανύμει χθε είναι δύο θέματα όπου υπάρχουν τροποποιήσεις. Πρόκειται για την τροπολογία 38 και 40. Για την 38 στον κατάλογο ψηφοφορίας υπάρχει ένα πλή, υπήρχε ένα πλήν, τώρα είναι ένα συν. Κυρία Μπιλμπάου, μια στιγμή επειδή είναι πολύ πολύπλοκο αυτό ο κατάλογος, καλύτερα όταν φτάσουμε στο συγκεκριμένο σημείο να σηκώσετε το χέρι σα, θα σα δώσω το λόγο για να απαντήσετε. Αλλιώ με τόσε τροπολογίε χάνουμε τον μπούσουλα και τον ίδιο τον γάβρο εξάλλου. Λοιπόν, θα μου, θα μου ζητήσετε το λόγο και θα εξηγήσετε περί τίνο πρόκειται. <clears throat> Ωραία. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία. Ναι, ναι. Ε, Τροπολογία 23 η Τουργάη Σάγκολο έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 2 λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία. Της εισηγητρίας είναι η τροπολογία 2. Πέρας. 18 ψήφισαν. 19 ψήφισαν, 12 υπέρ, 4 κατά και μία αποχή. Εγκρίνεται. Στη συνέχεια, η τροπολογία 24 του κυρίου Ασένη άρχεται η ψηφοφορία. Σε cierra la Πέρας 18 ψήφισαν, 18 υπέρ εγκρίνεται. Τροπολογία 3 εκπίπτει και περάμε στην 25 του κ. Ασένη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 18 ψήφισαν, όλοι υπέρ εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 26. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρα στις ψηφοφορίες. Δεκαεφτά ψήφισαν, όλοι υπέρ, εγκρίνεται. Η τροπολογία 29 άρχεται η ψηφοφορία για την 29. Άρχεται η ψηφοφορία λοιπόν για την τροπολογία 29. Πέρας. Απορρίπτεται. A ver, eh, se 14 ψήφοι κατά απορρίπτεται κατά συνέπεια. Επαναλαμβάνεται η τροπολογία για την 29. Ε, αν δεν, αν δεν έχετε κάρτα να σηκώνετε το χέρι σας παρακαλώ και να λέτε τι ψηφίζετε. Σε cierra la 18 ψήφισαν, 4 4-5, 14 κατά, Απορρίπτω την τροπολογία αυτή. Πάμε στην 27. Η Τούργα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ήθελα να αποσύρω την ε, τροπολογία αυτή, αλλά δεν πρόλαβα. Θέλω να ανακοινώσω την πρόθεσή μου να αποσύρω την ε, τροπολογία αυτή. Δεν είχαμε το χρόνο όμω να το κάνουμε. Ωραία, οπότε ψηφίζουμε την τροπολογία 27. <clears throat> Πέρας ψηφοφορία. 18 ψήφισαν, 7 υπέρ και 10 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 της εισηγήτριας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 11 υπέρ, 7 κατά, 18 ψήφισε συνολικά. Εγκρίνεται η τροπολογία. τροπολογία 31 του κυρίου Ιτουργάη. Πέρας ψηφοφορίας. 18 ψήφισαν, 7 υπέρ, 11 κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 10 της εισηγήτριας λέει. la enmienda, perdón, la enmienda La enmienda 30 ha sido retirada. Συγγνώμη, η τροπολογία 30 έχει αποσυρθεί, λέει. Όχι, όχι, πρέπει να ψηφίσουμε την 30, η οποία δεν έχει εκπέσει, λέει η πρόεδρο. 30 τη συζήτηση δεν έχει εκπέσει, λέει η πρόεδρος. Αρχίζουμε την ψηφοφορία στην τροπολογία 30, λέει η πρόεδρος. 8 υπέρ, 7 κατά. Εγκρίνεται η τροπολογία 30. Η 5 έχει αποσύρθει. Η τροπολογία 32 <clears throat> ως προσθήκη θα δώσει ψηφοφορία. Υπάρχει την ψηφοφορία. Λήξεις. 11 υπέρ 8 κατά εγκρίνεται. Η τροπολογία 6 τώρα. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μονάχα ήθελα να πω ότι εδώ υπάρχει μια προφορική τροποποίηση. Αλλάξαμε την αναφορά στις ε, εθνικές και περιφερειακές αρχές των κρατών μελών που ήταν οι αρμόδιες και λέμε απλώς οι αρμόδιες αρχές. Εντάξει, με αυτή την τροποποίηση άρχεται η ψηφοφορία της τροπολογίας παριθμών 6. Λίγη ψηφοφορία. 18 ψήφισαν όλοι υπέρ. Εγκρίνεται λοιπόν η τροπολογία υπερθυμών 6. Τροπολογία 33 του κύριου Ιτουργκάιθ. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. 12 υπέρ, 7 κατά εγκρίνεται. Εκπίπτει κατά συνέπεια τροπολογία 7 της εισηγήτριας. Περνάμε στην τροπολογία 34 η Τουργάη Αγγούλο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 14 υπέρ κατά 6 μονάχα, <coughs> επομένως εγκρίνεται και 34. Εκπίπτει τώρα η τροπολογία παριθμών 8 της εισηγήτριας. Περνάμε στην τροπολογία 9 της εισηγήτριας. Ε, Μου λέει η γραμματεία ότι υπάρχει μία παραπάνω ψήφο από την φιλελεύθερη ομάδα γιατί είναι τρει οι, οι των φιλελευθέρων και ψηφίζουν τέσσερι ένα από του φιλελεύθερου δεν πρέπει να ψηφίζει. Σα παρακαλώ να ελέγξετε. Είμαι αναπληρωματική. Είναι θέμα της ομάδας σας, δεν είναι δικό σας πρόβλημα. Εμεί σα λέμε ότι στη φιλελεύθερη ομάδα ψηφίζει ένα άτομο παραπάνω, επομένω κάποιο από του φιλελεύθερου πρέπει να σταματήσει να ψηφίζει, όχι εσεί κατά ανάγκη. Ο κύριο Γκάλερ δεν θα ψηφίζει λοιπόν. Περνάμε. Στην τροπολογία 9 της εισηγήτριας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 7 ψήφοι υπέρ, 9 κατά απορρίπτεται η τροπολογία 9 τη εισηγήτριας. επομένω περνάμε στην τροπολογία 35 Αρσένη. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 15 ψήφοι υπέρ, 2 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10 της εισηγήτριας και έτσι δίνω το λόγο για να εξηγήσει την ε, πρότασή της συμβαστική. Μάλιστα κυρία Πρόεδρε, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, αντί να λέμε οι κρατικές και περιφερειακές αρχές των κρατών μελών, λέμε απλώς οι αρμόδιες αρχές. Εντάξει. <clears throat> Με αυτή την τροποποίηση ψηφίζουμε την τροπολογία 10 της εισηγήτριας. Αρχή η ψηφοφορία. Πέρας. 19 <clears throat> ψήφισαν όλοι υπέρ. Εγκρίνεται η 10. Η τροπολογία 11 έχει αποσυρθεί. Οι τροπολογίες 36 και 37 που είναι ταυτόσιμες θέτω σε ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνονται 17 ψήφοι υπέρ, 3 κατά. Τροπολογία 38 τώρα. Η Άγγουλο, άρχεται η ψηφοφορία. Συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, εδώ ήθελα να σας υπενθυμίσω, όπως είχα πει στην αρχή. Στον κατάλογο ψηφοφορίας εμφανίζεται αρνητική σύσταση της συγγήτριας, αλλά θέλω να την υποστηρίξω αυτή την τροπολογία, θέλω να βάλω ένα σύνεκι. Εντάξει, αρχίζει και πάλι η ψηφοφορία για την 38, λέει η Πρόεδρος. Πέρας. Όχι, όχι, όχι, συγγνώμη λοιπόν. 9 υπέρ, 9 κατά, απορρίπτεται. Ακολουθεί τροπολογία 39, <clears throat> Αντζές Μπαρέα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 6 υπέρ, 14 κατά. Περνάμε στην τροπολογία 12 της εισηγήτριας άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 14 πέρα 6 κατά εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 13 της εισηγήτριας άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 14 υπέρ 6 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 14 της εισηγήτριας, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. 20 ψήφοι υπέρ, καμία ψηφός κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 40, η Τουργκάη Σάγκουλο, άρχεται η ψηφοφορία. Κυρία Πρόεδρε, και εδώ στον κατάλογο πρέπει να σας πω, προηγουμένως είχα ένα συν στον κατάλογο ψηφοφορίας, αλλά τώρα δεν την υποστηρίζω, έχει μείον κανονικά. Λοιπόν, ε, εξ αρχής ψηφοφορία για τις 40, λέει πρόεδρος. Πέρας. 10 ψήφοι υπέρ, 8 κατά, εγκρίνεται η τροπολογία 40. Τροπολογία 15, άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 20 ψήφοι υπέρ, καμία κατά, καμία αποχή, εγκρίνεται. 16 συζυγήτριας. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 6 ψήφοι υπέρ, 13 κατά. 41, αντρέ Μπαρέα. Άρχεται η ψηφοφορία. 17 την ψηφίσαμε, όχι την ψηφίσαμε. Νομίζω ότι εγκρίναμε τη 17. Λοιπόν, ας κάνουμε τη ψηφοφορία για τη 17. αρχή την ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίες. Εγκρίνεται 11 ψήφοι υπέρ, 8 κατά. Πάμε στην 41. Ανδρέας Μπαρέα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας τις ψηφοφορίες. Απορρίπτεται 14 ψήφοι κατά 5 ψήφοι υπέρ. Τροπολογία 18. Η Τουργκάης. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται 9 υπέρ 12 κατά. Η τροπολογία, η 19 έχει αποσυρθεί, πάμε στην τροπολογία 20 guys Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 12 ψηφί υπέρ 9 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22 ασένης Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 20 ψηφί καμία κατά. Η ένα έχει αποσυρθεί και η τροπολογία έχει εκπέσει. Θέλω να συγχαρώ λοιπόν την εισηγήτρια και έχει τελειώσει η ψήφος προσανατολισμού. Περνάμε στην έκθεση του κύριου Γκάλεχερ. Eh, Κύριε Γκάλαχερ, θέλετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ψηφίζουμε και τα τρία πλήρη μέλη. Σε σχέση με αυτό, αυτό που συμβαίνει είναι ότι χωρίζουμε την περιοχή αυτή του κόλπου από το υπόλοιπο γιατί είναι το ίδιο απόθυμα που μας συμβούλευσαν οι επιστήμονες. Και αν δεν το κάνουμε αυτό θα ήταν εντελώς αντίθετο με την κάλπ. Πρέπει να είμαστε συνεπείς. Ουσιαστικά αυτό είναι το, το πρόβλημα για όλες τις τροπολογίες και οι μερικές τροπολογίες μπορώ να τις δεχτώ. la derecha? ¿Cuál es? Ah. Bueno, pues eh, comenzamos la votación. Eh, a ver, en primer lugar, someto... Πρώτα απ' όλα, τροπολογία 19 του κυρίου Φερέιρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 20 ψήφοι κατά καμία υπέρ. Απορρίπτεται η 19. Συνεχίζουμε με 20, Αντρές Παρέα. Α, η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 18 ψηφίπερ, υπέρ, 2 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 21 Φερέρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται 6 ψήφοι υπέρ, 14 κατά. τον εισηγητή τώρα για μια προφορική τροπολογία στο άρθρο 5. Κύριε εισηγητά. Uh, Πρόεδρε, απλά θέλουμε να αντικαταστήσουμε την ε, αναφορά στο άρθρο 20 του κανονισμού 2371-2002 με το άρθρο 43.3 της ε, Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ψηφίζουμε τροπολογία 1 με την ε, με τις ευκρινήσεις του εισηγητή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 19 ψήφοι υπέρ καμία κατά. ψηφοφορία της τροπολογίας 22 της κυρίας Μπιλμπάου. Άρχεται η ψηφοφορία. Δεν μπόρεσα να ψηφίσω. Δεν δούλεψε το μαραφέτη μου λέει ο κύριος Παντήλια. Αρχίζει και πάλι η ψηφοφορία για την τροπολογία 22. Κυρία Μπιλμπάου, έχετε το λόγο, ναι. Στην τροποποίηση αυτή θέλω να αντικατοπτρίσω το εξής. Δεν αντικαθιστούμε το σημείο 2 του αρχικού κειμένου. Προσθέτουμε μονάχα ένα κομμάτι, χωρίς ε, μικρόφωνο η πρόοδος. Χωρίς μικρόφωνο η πρόοδος. Χωρίς μικρόφωνο η πρόοδος. Περνάμε στην τροπολογία Τρία τη συζήτρια, λέει η πρόεδρο, Έχει αποσυρθεί 23 προηγουμένω. ναι. Τρία της συζήτρια του εισηγητή, άρχεται η ψηφοφορία, λίγη ψηφοφορία. 18 υπέρ 2 κατά Ξεπερνάμε. Μάλλον δίνω το λόγο στον εισηγητή για μια προφορική τροποποίηση, την τροπολογία 2 που αντικαθιστά την 4. Έχετε το λόγο κύριε Γκάλαχερ. Thank you, Chair. And... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για αντικατάσταση του σημείου που αναφέρεται στις νέες αξίες για τα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 43 της ε, Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψηφίσουμε λοιπόν για τη 2, άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. 18-0 εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 5 του εισηγητή αυτή την ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 20 ψήφοι υπέρ, καμία κατά. Περνάμε στις τροπολογίες 25 και 24 που είναι ταυτόσιμες του εισηγητή και της κυρίας Μπιλμπάου. Κυρία Μπιλμπάου. Απλώς και μόνο να σας πω ότι εδώ χρειάζεται να υπάρχει μία αναφορά στον ε, νέο κανονισμό του Συμβουλίου και όχι τον 1627 όπως λέει η τροπολογία. Ωραία, με αυτή την προφορική τροποποίηση άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. 20 υπέρ κανείς κατά, εγκρίνεται κατά συνέπεια. Περνάμε <clears throat> το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 24 Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ε, ψηφοφορίας απορρίπτεται με ισοψηφία 10-10. Περνάμε στην τροπολογία 7 του εισηγητή. Άρχεται η ψηφοφορία. λήξης 18 <clears throat> ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8 του εισηγητή. Παρακαλώ, κύριε Ρόβιτς. Απλώς θέλω να ψηφίσω θετικά σε αυτή την περίπτωση γιατί δεν λειτουργήσε το μηχάνημά μου. Εντάξει, δεν αλλάζει το αποτέλεσμα έτσι κι αλλιώς, η πλειοψηφία ήταν υπέρ καταγράφουμε αυτό το οποίο είπατε. Περνάμε στην τροπολογία 8 του εισηγητή. Άρχεται η ψηφοφορία. Κλείνει η ψηφοφορία. 20 υπέρ κανείς κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 9 διαγραφής του εισηγητή άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 18 υπέρ 2 κατά. Η τροπολογία 10 του εισηγητή. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 20 υπέρ, κανείς κατά. Τροπολογία 27 του εισηγητή. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται πάλι με την ίδια, ψηφοφο... πλειοψηφία 20 υπέρ κανείς κατά. Τροπολογία 12 του εισηγητή. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται 17 υπέρ 2 κατά. Τροπολογία 10. Ε, Τη 12 την ψηφίσαμε. Η 28 εκπίπτει. Πάμε στη 13 του εισηγητή. Άρχεται την ψηφοφορία για τη 13. Πέρας. Απορρίπτεται 11 κατά 9 υπέρ. Τροπολογία 29 του εισηγητή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 20 υπέρ καμία ψήφος κατά. Τροπολογία 1 του εισηγητή. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 20 υπέρ κανείς κατά. Εγκρίνεται. Η 14 έχει εκπέσει. Τροπολογία 15, ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 15 υπέρ, 5 κατά εγκρίνεται. Η τροπολογία 15. Πάμε στην 2 του εισηγητή, άρχεται ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. 20 υπέρ, κανείς κατά εγκρίνεται. Η τροπολογία 16 είναι συμβατή. Την ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για τη 16. Πέρας. 18 υπέρ 2 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 17 της κυρίας Μπιλμπάου. Εξέπεσε μάλιστα. Και η 18 εξέπεσε. Η 18 δεν εξέπεσε. Ψηφίζουμε 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 14 ψήφοι υπέρ, πέντε κατά. <clears throat> Εγκρίνεται, συγχαίρω τον συγητή, δεν υπάρχει τελική ψηφοφορία βέβαια. Για την ψηφοφορία ανατολισμού και έτσι έχουμε τελειώσει τις ψηφοφορίες. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημέρας διάταξης. Δικό μου σφάλμα, αλλά η τροπολογία 17 εξέπιπτε αν θα ενεκρίνει το 19, η οποία δεν ενεκρίθη βέβαια. Νομίζω πρέπει να είχαμε ψηφίσει 17 λοιπόν, λέει η κυρία Μπιλμπάου. 24 ah, no, no. απερίφθη, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα κυρία Μπιλμπάου για τη 17. Εφόσον απερίφθη 24, εκπίπτει 17. Μα το πρώτο τμήμα της 24 δεν εκρήθη, λέει κυρία Μπιλμπάου. Αλλά το τμήμα το οποίο είναι ασύμβατο είναι το δεύτερο τμήμα της 24, οπότε Καλό, καλό να το διευκρινίσουμε. Πολύ καλά. Πολύ καλά κάνουμε. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημέρας της λοιπόν μετά από όλες αυτές τις περιπέτειες. Που είναι το θέμα του ΙΚΑΤ, του Διεθνούς Φορέα για τον Τόνο. Όπως ξέρετε, στο Ρεσίφε στη Βραζιλία θα λάβει χώρα η 21η συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής για την Προστασία του Τόνου του Ατλαντικού έγινε μάλλον. Ήταν δύο βουλευτές παρόντες, ο κύριος Ρωμέβα Ιρουέδα και εγώ η ίδια. Ζητήσαμε να είναι παρούσα και η Κομισιόν για να μας πληροφορήσει για τα πορίσματα και τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο RSCFER στη διάρκεια αυτής της ε, ετήσιας συνεδρίασης και καταρχήν, εάν συμφωνείτε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στους βουλευτές οι οποίοι θέλουν να πούνε κάτι και ήταν τμήμα της ε, αντιπροσωπείας ο κύριος Ρωμέβα συγκεκριμένα και μετά θέλω να κάνω και εγώ κάποια σύντομα σχόλια σε σχέση με τη συνεδρίαση αυτή τη ΕΚΑΤ και μετά θα δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν ώστε να μας εξηγήσει τη δική τους άποψη. Κύριε Ρωμέβα, προτιμάτε να μιλήσει πρώτα η Κομισιόν ή Κομισιόν, Κομισιόν. Είναι παρούσα η Κομισιόν και εγώ θα μιλήσω μετά την Κομισιόν. Έχετε το λόγο. Κύριο Δημό έχει το λόγο από την πλευρά τη Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Με δύο λόγια τα απορίσματα αυτής της αιτήσιας τακτικής συνεδρίασης. Η Κομισιόν σας παρουσίασε τις προσδοκίες και τους στόχους της Ένωσης για τη συνεδρίαση αυτή. Σήμερα ο απολογισμός είναι ικανοποιητικός. Καταρχήν θέματα που δεν είναι θέματα κόκκινου τόνου. Γιατί ορισμένοι έδωσαν λιγότερη προσοχή σε άλλα θέματα που είναι εξίσου σημαντικά. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες θεμάτων που συζητήθηκαν εκεί στη Βραζιλία, στην ΙΚΑΤ. Πρώτον, η τήρηση των υποχρεώσεων, compliance, αγγλικά. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και για την Ένωση και για τον ΚΑΤ. Δηλαδή, εμβάθυνση της διαδικασίας. Το Μάρτιο είχαμε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Εφαρμογής στη Βαρκελόνη. Ο απολογισμός θετικός στην ΕΚΑΤ όσον αφορά την compliance. Η διαδικασία ελέγχου τήρησης των υποχρεώσεων των συμβαλωμένων μερών που υπάρχουν δυσκολίες που υπάρχουν τα κενά με επιστολή προσπάθεια να διορθωθούν αυτά τα προβλήματα και να βγουν και τα συμπεράσματα. Στην ετήσια συνεδρίαση της ΕΚΑΤ άρχισε να ισχύει ένα σύστημα κυρώσεων για χώρες που δεν πληρούν τις υποχρεώσεις σε σύστημα που πρότεινε η Ένωση και που εμπνέεται από τον κανονισμό ελέγχου της Ένωσης, τον πρόσφατο. Δεύτερο στοιχείο είναι τα μεγάλα αποθέματα για τον τόνο, για τον ξηφία του Ατλαντικού, τον ξηφία της Μεσογείου και άλλα είδη. Η Ένωση στηρίζεται στην επιστημονική, στην επιστημονικά δεδομένα. Η Επιστημονική Επιτροπή του ΕΚΑΤ είχε κάνει συστάσεις να μειωθεί το επίπεδο των ΤΑΚ. Με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι μειώθηκε το ΤΑΚ Οπότε η Ένωση προσπάθησε να υπερασπίσει τα συμφέροντα του στόλου της. Ο απολογισμό είναι ικανοποιητικό. Δηλαδή η επιστημονική γνωμοδότηση τηρήθηκε και η Ένωση, τα συμφέροντα μάλλον της Ένωσης, προασπίστηκαν. Το απόθυμα του ξηφία του Βόρειο Ατλαντικού που είχε δυσκολίες μετά από 10 χρόνια προγράμματος δράσης του ΙΚΑΤ επανασυστήθηκε ο το απόθεμα με καλό επίπεδο ζωικής βιομάζας. Άρα θετικά τα αποτελέσματα και εδώ, της ΣΥΚΑΤ. Καρχαρίας. Όπως είπαμε η Ένωση ήθελε να προωθήσει την έγκριση μέτρων διατήρησης προστασίας του Καρχαρία. Δυστυχώς εδώ ο απολογισμός είναι μέτριος. Εγκρίθηκαν μεν μέτρα προστασίας του Καρχαρία Αλεπού και Ρενάχ που είναι τα πια ευάλωτα είδη πέρυσι δεν το είχαμε καταφέρει αυτό αλλά δεν καταφέραμε να εγκριθούν άλλες προτάσεις για τον Καρχαρία αυτό, σε αυτό θα επανέλθουμε δυστυχώς αυτή τη φορά δεν καταφέραμε να πετύχουμε συνένεση για τα μέτρα αυτά για την προστασία του Καρχαρία Επίσης υπήρχαν και μέτρα προστασίας των πτηνών της θάλασσας. Εδώ, για άλλους λόγους, δεν καταφέραμε να εγκριθούν συμπληρωματικά μέτρα για την προστασία τους. Ερχόμαστε τώρα στον κόκκινο τόνο, που ήταν το κύριο θέμα. Σε σχέση με τους στόχους της Ένωσης, ο απολογισμός μας είναι θετικός, ικανοποιητικός τα κύρια μέτρα που εγκρίθηκαν σημαίνουν σημαντικές θυσίες για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Ωστόσο οι θυσίες αυτές ήταν αναγκαίες προκειμένου να έχουμε διατήρηση του αποθέματος του κόκκινου τόνου. Τα κύρια μέτρα είναι μεγάλη μείωση του ΤΑΚ. Περάμε από 22.000 τόνους σε 13.700. Η επιστημονική γνωμοδότηση πάλι για ΤΑΚ μεταξύ 8.500 και 15.000 τηρήθηκε. Δεύτερον, η εποχή αλίας μειώθηκε στο μισό για το γρηγρία. Δηλαδή από τα μέσα Μαΐου μέχρι τα μέσα Ιουνίου για τα γρηγρία. Καμία άλλη ευελιξία μετά τις 15 Ιουνίου. Τρίτο στοιχείο πολύ σημαντικό, το υπερβάλλον δυναμικό του στόλου. Όπως θυμόσαστε, η Ένωση στη συνεδρία αυτή πήγε με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα μείωσης του δυναμικού της Ένωσης. Πετύχαμε αντίστοιχες προσπάθειες και από τις άλλες χώρες. Θετικό αυτό. Δηλαδή πρόγραμμα μείωσης του στόλου. Δεσμευτικό. Εγκρίθηκε. Διότι το υπερβάλλον δυναμικό του στόλου για τον κόκκινο τόνο ήταν μια μείζων συνιστόσα για την υπεραλίευση του τόνου αυτού. Ένα τελευταίο στοιχείο, τα έγγραφα αλλιευμάτων. λέτε αυτό στο εμπόριο διεθνώς. Η ΕΚΑΤ τα τελευταία χρόνια ε, εισήγαγε ένα σύστημα πιστοποίησης για να υπάρχει η του, του τόνου από την αλλίευσή του μέχρι την τελική κατανάλωση ασχοληθήκαμε και πάλι με το έγγραφο αυτό και ενισχύθηκε το σύστημα. Αυτά με δύο λόγια ήταν κύρια στοιχεία αυτής της ετήσιας συνεδρίασης. Για την Ένωση είναι ικανοποιητικά. Σημαίνουν προσπάθειες και θυσίες και για τα κρατημέλη και για τον κοινωνικό στόλο, αλλά οι θυσίες αυτές ήταν αναγκαίες. Πρώτον να τηρούνται οι επιστημονικές προτάσεις και δεύτερον η διατήρηση του αποθέματος του τόνου. Η ΙΚΑΤ απέδειξε ότι και μπορεί να διαχειρίζεται το σύνολο των αποθεμάτων και δεύτερον απέδειξε ότι είναι στο ύψος της ευθύνη της. Όλα τα μέτρα εγκρίθηκαν με συνένεση από τα 48 συμβαλόμενα μέρη. Αυτό είναι ένα σαφές σινιάλο και για τη δέσμευση εφαρμογής των υποχρεώσεων και για μια πολιτική βούληση που λέει ότι η ΕΚΑΤ μπορεί να παίξει το ρόλο και την εντολή που της έχει δοθεί. Eh, Ευχαριστώ κύριε Ρομέβα. Θέλετε να λάβετε το λόγο. Προηγουμένως θα ήθελα να σας πω το εξή. Στις 10.30 ξεκινάει η ακρόαση για την κοινή αλληλευτική πολιτική. Έχετε και εσείς ένα σημείο στη μέση διάταξη. Έχετε κάθε συμφέρον λοιπόν να είσαστε σύντομο, σα, το λέω, αστειευωμένοι βέβαια. Esto cuánto tiempo me da, pregunto, para calcular. Πόσο χρόνο έχω, παρακαλώ. Λίγο, λίγο, λέει η Πολύ λίγο. Eh, λοιπόν, πέντε τηλεγραφικέ φράσει. Κύριε Ρωμέβα. Δεν ακούγονται τα αγγλικά. Υπάρχει... Υπάρχουν παρεμβολές. Το μικρόφωνο μου φταίει ή κάποιος άλλος φταίει. Κάποιος έχει ανοιχτό το τηλέφωνο του, λέει ο κύριος Στίβενσον for example, with my... It's better now. Somebody's mobile. Eh, you, you are okay now? It's okay. okay, venga, señor Romeva. Πάμε κύριε Ρομέβα. Σας το λέω τηλεγραφικά λοιπόν σε πέντε σημεία μονάχα. Πρώτον, έχοντας παρακολουθήσει όλη τη, διαδικα... όλη τη διαδικασία της συνεδρίασης της ΙΚΑΤ από την αρχή ως το τέλος, σε εννέα μέρες στο Ρεσίφε, Είμαι λιγότερο αισιόδοξο από την Κομισιόν. Νομίζω ότι είναι κάπως λεπτή η θέση της ΙΚΑΤ σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία της, όσο και επίσης σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των προτάσεών της. Και αυτό γιατί έχω να σας παρουσιάσω μια σειρά από επιχειρήματα υπέρ αυτής της ε, θέσης. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία μεταφέρονται από το ένα χρόνο στον άλλο χωρίς λήψη απόφαση. Ήμουν στο Μαρακές πέρσι που ήταν η προηγούμενη συνεδρία της ΕΚΑΤ. Εφέτος επιβεβαιώθηκε ακριβώς η ίδια κατάσταση. Είναι απαραίτητο να σκεφτούμε καλύτερα ποιο είναι ο ρόλο και η αποτελεσματικότητα ενό φορέα όπω για να αντιμετωπίσει την κύρια πρόκληση που είναι η ανάκαμψη των αλληλευτικών στόκ. Πάρα πολύ σύντομα λοιπόν. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη συμμόρφωση, compliance. Δύο σκέψεις εδώ θέλω να σας κάνω. Είναι γεγονός ότι όλο και περισσότερες πληροφορίες έχουμε, όλο και περισσότερη ικανότητα έχουμε να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση των κανόνων, είναι παράλληλα γεγονός ότι η εντύπωση που έχω για την ΙΚΑΤ είναι ότι υπάρχει μια σιωπηρή συμφωνία να αλληλοκαλύπτονται οι ε, κακές πρακτικές που κάνουν τα κράτη-μέλη. Κανείς δεν καταγγέλει κανένα και λέμε ότι εγώ δεν σε καταγγέλω, σε λέμε καταγγέλλεις και έτσι υπάρχει μια αλληλοπροστασία. Αυτή είναι μια γενική εικόνα, ήταν θλιβερό. Θλιβερή αυτή η εικόνα γιατί οδηγεί και σε αντικά αποτελέσματα, κάτι το οποίο δεν ανέφερε η Κομισιόν. Σαν παράδειγμα ήταν συζήτηση που είχαμε σε σχέση με τα παρασυρώμενα δίκτυα του Μαρόκου. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο το έχουμε θέσει πολλές φορές στην Επιτροπή μας πολλοί για την χρήση παρασυρωμένων δικτύων από το Μαρόκο Υπάρχει υποχρέωση από την πλευρά του Μαρόκου να καταργήσει τη χρήση αυτού του είδους παρασυρωμένων δικτύων με απόφαση όχι μόνο τη ΣΥΚΑΤ αλλά και γιατί παίρνει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνει αυτή την κατάργηση των παρασυρωμένων δικτύων εμείς διαπιστώνουμε ότι αυτό δεν έγινε στην πραγματικότητα και στην ΙΚΑΤ έλαβε χώρα μια συζήτηση για το πώς να δικαιολογηθεί η μη συμμόρφωση του Μαρόκου για την <clears throat> εξάλληψη αυτών των δικτύων, αυτό οδηγεί σε πραγματική αμφιβολία αν εφαρμόζονται οι κανόνες της ΙΚΑΤ ή δίνονται σιωπηρέ παρεκκλήσεις, όπως στην περίπτωση του Μαρόκου. Το Μαρόκο ζήτησε μια εξαίρεση, κανείς δεν ήταν κατά αυτής της εξαίρεσης, επομένως σιωπηρά απεδέχθησαν τα υπόλοιπα συμβαλόμενα κράτη-μέλη αυτή την εξαίρεση. Η συνεδρίαση του Ρεσίφε είχε σαν πρόθεση να επισημοποιήσει αυτή την εξαίρεση και να την κάνει όχι μόνο χασιοπηρή αλλά εκπεφρασμένη. Αλλά αυτό δεν είναι ο πιο νομότυπος τρόπος, ούτε καν ο πιο νόμιμος τρόπος να κάνουμε πράγματα. Και ουσιαστικά έρουμε έτσι την υποχρέωση του Μαρόκου να καταργήσει τα παρασυρώμενα δίκτυα, τα οποία θίγουν όχι μονάχα την αλία στην περιοχή του Μαρόκου, αλλά και σε άλλες περιοχές του Νοτιού Ατλαντικού, όπου αλλιεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο σημείο. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στις συνεδριάσεις της ΕΚΑΤ. Το είπε και η Κομισιόν ότι υπήρξε ένα πρόβλημα χρόνου. Υπήρξε πρόβλημα χρόνου γιατί δεν ήταν σαφείς και οι προτεραιότητε. Είχαμε εννέα ημέρες. Μέσα σε αυτές τις εννέα μέρε έλαβαν χώρα πάρα πολύ εντατικέ συνεδριάσεις. Και αυτό το οποίο γινόταν ήταν κάθε φορά πετούσαμε το μπαλάκι για την επόμενη μέρα. Αναβάλαμε, αναβάλαμε, αναβάλαμε, αναβάλαμε και όταν φτάναμε στο ουσιαστικό κομμάτι των συζητήσεων δεν είχαμε το χρόνο να συζητήσουμε ορισμένα από τα θέματα τα οποία είχαν συζητηθεί προηγουμένω και επομένω για θέματα όπω ήταν τα καρχαριοειδή, όπω είναι τα θαλάσσια πτηνά, οι κορμοράνοι, οι χελώνε, όλα αυτά τα θέματα δεν μπορέσαμε να τα συζητήσουμε επαρκώ. Αυτό ήταν διαρθρωτική αστοχία στη σε αυτή τη ΣΥΚΑΤ. Είναι γεγονό ότι ο γαλαζόπτερο ή ερυθρό τόνο ήταν το κύριο θέμα τη ε, συνεδρία τη ΣΥΚΑΤ, αλλά δεν μπορούμε κάθε φορά να αναβάλουμε για τον επόμενο χρόνο τη λήψη αποφάσεων οι οποίες είναι σημαντικές και που με τον τρόπο αυτό υποσκάπτουμε την αξιοπιστία της ΙΤΑΤ. Τρίτο σημείο. Όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αλλά και σε ό,τι αφορά το αποτέλεσμα είναι ο ερυθρός τόνος. Ο ερυθρός τόνος ήταν το αστέρι αυτών των συζητήσεων, ήταν το κέντρο όλων των συνεδριάσεων και σε μεγάλο βαθμό επηρέασε και τις αποφάσεις σε σχέση με άλλα αλλιεύματα και σε άλλα θέματα. Θέλω εδώ να αναφερθώ στο θέμα της ερμηνείας των αποφάσεων που έλειψαν από την ΙΚΑΤ. Όλοι μας συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα. Ούτε καν οι επιστήμονες δεν είναι σίγουροι. Βρισκόμαστε πάντα στο τομέα, στον τομέα των πιθανότητων. Υπάρχουν πιθανότητες να αυξηθούν τα στόκ, πιθανότητες να καταρρεύσουν τα αλλιευτικά στόκ του ερυθρού τόχου. Επομένως, το πραγματικό ερώτημα είναι τι επίπεδο κινδύνου μπορούμε να αποδεχτούμε βασιζόμενοι σε αυτές τις πιθανότητες. Και εδώ διαφωνώ για το ότι το γεγονός ότι αποφασίστηκε να υπάρξει το όριο των 8.000 τόνων ήταν σωστό. Οι πιθανότητες που μας δώσαν οι επιστήμονες, όχι μονάχα στη συνεδρίαση του Ρεσίφ, αλλά και στη Μαδρίτη πριν από μερικές μέρες σε μια συνεδρίαση η οποία ήταν μονογραφική σε σχέση με την κατάσταση του, των αλλιευμάτων του ερυθρού τόνου, το 8.000 τόνοι σημαίνει ο κίνδυνο 50% να μην υπάρξει ανάκαμψη των αποθεμάτων ερυθρού τόνου. Επομένως όλα αυτά δεν μας εξασφαλίζουν μια αποτελεσματικότητα στον τομέα αυτό. Επίσης σε όλη αυτή τη διαδικασία ετέθη επιτάπτως κάτι το οποίο για μένα ήταν αποφασιστικό και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με ειδικό τρόπο στο επόμενο χρονικό διάστημα που ήταν η διαπίστωση ότι υπάρχουν συγκυρίες που πρέπει να μας οδηγήσουν να συμπεριλάβουμε τον τόνο στο παράτημα 1 της ΣΥΤΕΣ, επειδή ακριβώς υπάρχει κίνδυνος να μην ανακάμψουν τα αλληλευτικά αποθέματα. Αν λοιπόν γίνει αυτή η συμπερίληψη του ερθρού τόνου στα προστατευόμενα είδη της ήτες στην Τόχα, αυτό είναι ένα προηγούμενο να έχουμε αλλιευτικά θαλάσσια είδη σε αυτόν τον κατάλογο. Αλλά η συζήτηση δεν έχει κλείσει, κατά την άποψή μου είναι πιο ανοιχτή παραποτέ και οι 8.000 τόνοι οι οποίοι έχουν εγκριθεί αυξάνουν κατά την άποψή μου αυτόν τον κίνδυνο μη ανάκαμψη των ε, αλλιευμάτων όταν έγινε η επιστημονική αξιολόγηση τονίστηκε ότι έπρεπε να γίνει μια αξιολόγηση επί τη βάση των τωρινών συνθήκων και όχι σε ένα πιθανολογικό σενάριο πιθανής ανάκαμψης. Τα τωρινά αλλιεύματα, αλλιευτικά στόκ είναι τέτοια που να θεωρηθεί ότι ο τόνος ο θα πρέπει να περιληφθεί στα προστατευόμενα είδη της ΙΤΕΣ. Για μένα λοιπόν το συμπέρασμα αυτό της ε, ΙΚΑΤ για 8.000 τόνους δεν είναι καλά νέα για να εξασφαλιστεί η ανάκαμψη των αλληλευτικών αποθεμάτων ερυθρού τόνου και ουσιαστικά ανοίγει μια συζήτηση για την προστασία του τόνου στην σύνδεση. Επίσης, <clears throat> τα έγγραφα για την αλίευση είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις σε σχέση με το περιεχόμενο αυτών των εγγράφων. Εγώ συμφωνώ ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία, και το λέω και πάλι, που είναι σημαντικές καιροτομίε. Καταρχήν, το ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση και να χρησιμοποιείται ένα σύστημα βαθμών ή μορίων που έχουμε προτείνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το οποίο το επικρότω γιατί είναι ένα καλύτερο τρόπο να ρυθμίσουμε τα θέματα αυτά. Και ένα δεύτερο σημείο το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και το λέω και τώρα, που είναι η υποχρέωση για μείωση τη αλληλευτική ικανότητα και αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο, πρέπει να το αναγνωρίσουμε, πρέπει να το καταγράψουμε. Και έρχομαι τώρα στο τρίτο σημείο που είναι τα έγγραφα αυτά για την ε, αλίευση έχουν βελτιωθεί γιατί είναι πιο διάφανα αυτά τα έγγραφα, αλλά είναι απαραίτητο να δούμε το εξής. Περιμένω να δω την τελική βέβαια μορφή των εγγράφων αυτών, αλλά υπήρξε μια σημαντική αίτηση για τα έγγραφα αυτά, για τα αλλιεύματα, να περιληφθούν στο σύνολο των πληροφοριών όλα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την αποθήκευση κατεψυγμένου τόνου μετά την αμβλίευση, γιατί αυτό είναι μια ειδική αίτηση του αλληλευτικού τομέα, γιατί θα μας επιτρέψει μια μεγαλύτερη ανιχνευσιμότητα της σύνολης διαδικασίας που ξεκινάει από την αλίευση του τόνου μέχρι την τελική πώληση του ερυθρού τόνου. Επομένως, <clears throat> είναι απαραίτητο να θέσουμε σοβαρά το θέμα αυτό της ε, προβληματικής σε σχέση με την ε, εντολή που θα πρέπει να δοθεί σε σχέση με τα έγγραφα αυτά αλίευσης. Αυτά. Eh, Ωραία. Και εγώ θέλω να κάνω μερικές ε, διευκρινήσεις και παρατηρήσεις σε σχέση με αυτά που είπαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές και ξεκινώ με τον ερυθρό τόνο. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έλαβε χώρα στο Ρεσίφε ήταν η μόνη δυνατή λύση η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί. Πολλέ φορέ στην περίπτωση τη αλίας δεν επιλέγεται ούτε η καλύτερη ούτε η χειρότερη λύση, αλλά απλώ η εφικτή λύση. Και τονίζω ότι αυτό ήταν πάντα μέσα στα πλαίσια των επιστημονικών εμπειρογνώμων των επιστημονικών ε, στοιχείων. Πάντα δουλεύουμε με πιθανότητες, δεν μπορούμε ποτέ να έχουμε βεβαιότητες. Επομένως πρέπει να χαράξουμε μια ε, μακροχρόνια στρατηγική και θεωρεί το σύνολο των επιστημόνων, οι επιστημονικές επιτροπές, ότι σε δύο χρόνια μπορούμε να έχουμε καλύτερες καταστάσεις. Και νομίζω ότι είναι καλύτερη λύση γιατί εάν λέγαμε ότι δεν θα υπάρξει καθόλου αλληλεία ερυθρού τόνου, αυτό θα σήμαινε ότι θα ανθούσε η παράνομη αλληλεία. Είναι πολύ ψηλή η τιμή του κρέατος του ερυθρού τόνου και αυτό σήμαινε ότι αν υπήρχε απαγόρευση θα γινόταν λαθρέα και μόνο. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι η λύση στην οποία καταλήξαμε ήταν η μόνη ρεαλιστική και εφικτή λύση. <clears throat> πιστεύω επίση ότι οι προσπάθειε που θα πρέπει να καταβληθούν από του στόλου που αλλιεύουν τον ε, ερυθρό τόνο θα πρέπει να είναι σημαντικέ. Θα αλλιεύουν μονάχα ένα μήνα το χρόνο. Είναι μείωση αλλιευτική ικανότητα 50% και νομίζω ότι αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική θυσία για τους αλίες του ερυθρού τόνου. Και υπενθυμίζω αυτά τα οποία ελέγχθηκαν ελέγχθηκαν στην Μαδρίτη θέσανε <clears throat> τρεις, τρία κριτήρια τα οποία είναι απόλυτα σαφή και το τρίτο αφορούσε την εφαρμογή των συνολικών αλλιευμάτων. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για συνολική απαγόρευση. Επομένως το πρόβλημά μας είναι με την Ιαπωνία. Η, Ιαπωνία είπε ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση να περιληφθεί ο ερυθρό τόνο στο παράτημα 1 τη ΣΥΤΕΣ και επειδή η Ιαπωνία είναι ο κύριο εισαγωγέα ερυθρού τόνου, καταλαβαίνετε ότι χωρί την Ιαπωνία δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ήταν απαραίτητο λοιπόν να έχουμε ένα ρεαλιστικό σχέδιο το οποίο δεν θα είχε μαξιμαλιστικό χαρακτήρα που δεν θα είχε κανένα θετικό αποτέλεσμα. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα τώρα στην Κομισιόν, <clears throat> όχι, για την όχι για τον, για τον ερυθρό τόνο, αλλά για άλλα είδη όπου έχουν τεθεί συνολικά αλλιεύματα μικρότερα από αυτά που έχει προτείνει η Επιστημονική Επιτροπή. Πρόκειται για είδη στα οποία δεν είναι σε δύσκολη κατάσταση. Γιατί δέχτηκε λοιπόν η Κομισιόν αυτή την ε, μείωση. Και έρχομαι στο θέμα των καρχαριδών. σε αυτά τα οποία αναφερθήκατε κι εσείς κύριε Ρωμέβα, ότι υπήρξε μια ευκαμψία, δεν είχαν εκπληρωθεί πλήρως οι υποχρεώσεις. Καθυστερούν προφανώς οι πολυμερείς οργανισμοί να καταλήξουν σε αποφάσεις και αυτό είναι λογικό γιατί έχουν πολλά συμβαλόμενα μέρη. Αν θυμάμαι καλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποβάλει μια πρόταση για το να μην εκφορτώνονται ε, οι σφυροκέφαλοι καρχαρίες. Αυτή ήταν η πρόταση αλλά <clears throat> εφέτος υπήρξε η απαγόρευση της ε, αλίας του σφυροκέφαλου Καρχαρή εκτός από, το, από την περίπτωση του Μεξικού όπου υπήρχε ένα πολιτικό πρόβλημα. Επίσης το θέμα των παρασυρωμένων δικτύων του Μαρόκου για την Ευρώπη, για τις ευρωπαϊκές χώρες αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο δράμα. Το γνωρίζουν οι Βρετανοί, το γνωρίζουν οι Ισπανοί, το γνωρίζουν και οι Ιρλανδοί. Πολλές φορές υπήρξε μια πολύ μεγάλη ε, διάκριση σε ό,τι αφορά την αλία στην ε, στη Μεσόγειο για την Παλαμίδα. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι το γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα και την προβληματική, ότι μέσα από την Αλευτική Συμφωνία με το Μαρόκο δόθηκαν χρήματα στο Μαρόκο για να καταργήσει την, την χρήση των παρασυρωμένων δικτύων. Αλλά παράλληλα γνωρίζετε ότι υπάρχει το πρόβλημα της παράνομης Πρέπει λοιπόν να δεχτούμε μερικές φορές τις πραγματικότητες. Πάντως, μετά από το 2011 είναι σαφές ότι δεν θα υπάρχει καμία απολύτως παρέκκληση σε ό,τι αφορά τα παρασυρώμενα δίκτυα και ίσως για πρώτη φορά να επιληθεί το θέμα αυτό. Θέλω να θέσω μια ακόμα ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι το θέμα του 15% ανοχής σε σχέση με το ελάχιστο μέγεθος των ε, ξηφιών στη Μεσόγειο που η Κομισιόν κατήργησε αυτό το στοιχείο. Θα να ξέρω για το 2010 τι ακριβώς θα κάνει η Κομισιόν με αυτό το περιθώριο ε, ανοχή σε σχέση με το μέγεθος του ξυφία στη Μεσόγειο. Γιατί του χρόνου θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση για αυτό το θέμα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι και εδώ η Επιστημονική Επιτροπή συμφώνησε για το γεγονός ότι είναι καλό να υπάρχει αυτή, αυτό το περιθώριο του 15% για να μπορούμε να παρακολουθήσουμε καλύτερα την εξέλιξη αυτών των αλληλευτικών πόρων. Τι θα γίνει όταν δεν θα υπάρχει αυτή η, η ανοχή και ποια θα είναι η άλλη η αντιμετώπιση από την πλευρά της Κομισιόν άλλων θεμάτων που δεν εμπίπτουν στα συνολικά αλλιεύματα. Πώς θα αντιμετωπίσετε λοιπόν τα θέματα αυτά των ανοχών στο μέγεθο των τόνων. Η, η κυρία Αντρέ Μπαρέα έχει το λόγο και μετά θα δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν. Αντρέ Μπαρέα. Πάρα πολύ σύντομα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα σε σχέση με την ε, εγκυρότητα των αποφάσεων ΕΚΑΤ Μπορεί κανείς να πει πολλά πράγματα για πολλές περιπτώσεις, αλλά τόνισε ο κύριος ε, Ρωμέβα ότι εξασφαλίστηκε να υπάρχει έλεγχος του, της πρόσβασης των αλευτικών στόλων, υπάρχει το σύστημα των βαθμών και υπάρχει και κάποια προστασία των αλλιευμάτων. Εγώ θέλω να θέσω τώρα ένα ερώτημα προς την Κομισιόν. Έχετε κάνει μια ειδική αξιολόγηση της παραδοσιακής ε, αλίας του ερυθρού τόνου στην ε, μεσογειακή, ε, στις μεσογειακές ακτές. Και όλα αυτά για να διατηρήσουμε την παραδοσιακή μορφή αλίας του τόνου. Eh, Παρακαλώ, έχει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους κοινοβουλευτικούς για τα ερωτήματά τους. Δεν θα απαντήσω ίσως σε όλα τα σημεία, αλλά θέλω να κάνω μερικές συγκεκριμένες παρατήρησεις. η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τα συνολικά αλλιεύματα ανταποκρίνεται στις προτάσεις Επιστημονικής Επιτροπής σε σχέση με τα συνολικά αλλιεύματα. Τώρα, τα τωρινά σχέδια διαχείρισης, <clears throat> αν υπολογίσουμε προσεκτικά τις ποσοστώσεις, δεν ανταποκρίνονται στα συνολικά αλλιεύματα. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει μια μείωση των ποσοστώσεων μετά την μείωση των ε, συνολικών αλλιευμάτων. Για τον Ξηφία στο Βόρειο Ατλαντικό, από μία πλευρά είναι μια επιτυχία της ΙΚΑΤ, έχουν ανακάμψει τα αποθέματα. Αλλά συγχρόνως η Επιστημονική Επιτροπή ζήτησε να μειωθούν τα συνολικά λίγματα. Είμαστε λοιπόν σε μια παράδοξη κατάσταση. Θέσαμε το ερώτημα στους επιστήμονες και μας είπαν ότι όταν έγινε η αξιολόγηση των αποθεμάτων εφέτος ε, αναθεωρήσανε μερικά από τα σενάριά τους σε σχέση με την παραγωγικότητα των ξηφιών. Γι' αυτό τον λόγο, από τη μία πλευρά είχαμε αυτή την επιτυχία ότι υπήρξε ανάκαμψη με των αποθεμάτων του ξηφία στο Βόρειο Ατλαντικό, αλλά συγχρόνω οι επιστήμονε ζητούν να αλλάξουμε λιγάκι τα σενάριά μα και να μειώσουμε ελαφρά τα συνολικά αλλιεύματα. Γι' αυτό καταλήξαμε να μειώσουμε τα αλλιεύματα και για τον ξηφία στο Βόρειο Ατλαντικό και στο Νότιο Ατλαντικό, ακολουθώντα τι προτάσει τη Επιστημονική Επιτροπή τη ΙΚΑΤ. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο τέθη αφορούσε το περιθώριο ανοχή για το μέγεθος του ψηφία, το οποίο συζητήθηκε στη συζήτηση της, στη συνεδρία της παραμένει μέσα στο πλαίσιο ανάκαμψης για τον ε, ξηφία του Ατλαντικού και είναι ένα σημείο το οποίο, όπως θυμόσαστε, αντιμετωπίστηκε στη συνεδρία για τα ΤΑΚ και τις ε, κότες της ε, ποσοστώσης πέρσι. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας ένα τέτοιο μέτρο δεν μπορεί να περιλαμβάνεται στον ετήσιο κανονισμό για τις δυνατότητες αλίας. Γι' αυτό ε, η Κομισιόν προετοιμάζεται να υποβάλει μια νέα πρόταση στον κανονισμό, ε, τον εκτελεστικό κανονισμό για τα μεγάλα μεταναστευτικά είδη ηχθείων, που θα περιλαμβάνει και τεχνικά μέσα και, τεχ... και τρόπους ελέγχους για την αλία ε, των τονοειδών και εκεί θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί και το θέμα του ξύφια. Τώρα, σε ό,τι αφορά την βιοτεχνική παραδοσιακή αλία του τόνου, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αποτέλεσε αντικείμενο ε, ιδιαίτερη συζήτηση στην ετήσια συνεδρίαση τη ΙΚΑΤ. Είναι ένα είδο αλίας όπου το επίπεδο ελέγχου θεωρείται ότι είναι επαρκές και φυσικά πρέπει να τηρούνται απόλυτα οι ποσοστώσεις και είναι ένα είδος αλίας το οποίο έχει μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον γιατί οι επιστήμονες επειδή είναι μια παραδοσιακή μορφή αλίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν επωφελώς τα στοιχεία τα οποία προέρχονται. Αλλά και πάλι σας λέω δεν έτυχε ιδιαίτερη μνήα σε αυτό το θέμα στην ετήσια συνεδρία στη Τσίκα. Τώρα θέλω να κάνω και ορισμένα σχόλια μετά από αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα που είπε ο κ. Ρωμέβα συμφωνώ απόλυτα μαζί του ότι δεν μπορούμε να αναβάλουμε στο δυναικές αποφάσεις για τα καρχαριοειδή. Για μας οι αποφάσεις που ελήφθησαν πράγματι δεν είναι ικανοποιητικέ. Πρέπει να ληφθούν και άλλα μέτρα και του χρόνου και πάλι θα πρέπει να πιέσουμε για την έγκριση μέτρων που θα εξασφαλίσουν την καλύτερη προστασία των καρχαριών. Αυτό είναι σημαντικό. Δεύτερον, για το θέμα τη συμμόρφωση, το σεβασμό των υποχρεώσεων. Εγώ θέλω να επιμείνω στο γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε σαφές ενώπιον όλων ποιο είναι το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες για την τήρηση των υποχρεώσεων. Ιδιαίτερα για τον ερυθρό τόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε ποια ήταν τα αποτελέσματα των ελέγχων και των επιθεωρήσεων στην ανοιχτή θάλασσα σε ό,τι αφορά την αλληλεία του ερυθρού τόνου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν κατέδειξε ποια ήταν τα πορίσματα αυτών των ελέγχων και είναι φανερό ότι η Ευρώπη έχει επενδύσει πολύ στον έλεγχο για την περίπτωση του ερθού τόνου. Έχει τεράστια μέσα τα οποία έθεσε σε χρήση για να υπάρξει έλεγχο στι αλλιέ και κατέληξε και στη συνεδρία τη ΙΚΑΤ ποια είναι τα προβλήματα και κα... κατέληξε και να δακτυλοδεικτήσει και τι χώρε οι οποίε δεν σέβονται τι υποχρεώσει του. Επίση για τα συνολικά αλλιεύματα ερυθρού τόνου έχουμε διάφορα επιστημονικά υποδείγματα τα οποία χρησιμοποιούνται και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προφανώς βασίζεται στις καλύτερες επιστημονικές εκθέσεις και πρόκειται συγκεκριμένα για τη θέση της Επιστημονικής Επιτροπής της ΙΚΑΤ όπως παρουσιάστηκε τον προηγούμενο Οκτώβρη και ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η έκθεση να υπάρχουν συνολικά αλλιεύματα μεταξύ 8 και 15.000 τόνων ε, τόνου. Εμείς λοιπόν ακολουθήσαμε αυτή την άποψη της ε, Επιστημονικής Επιτροπής ΙΚΑΤ σε σχέση με τα συνολικά λιεύματα. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα παρασυρώμενα δίκτυα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ιδιαίτερα στεναρή σε σχέση με το θέμα αυτό, τονίσαμε σαφώ και ζητήσαμε να καταγραφεί πλήρω στα πρακτικά το ότι δεν θα υπάρξει καμία δυνατή περαιτέρω παράταση της εξαίρεσης η οποία ισχύει για τον Μαρόκο. Από τη στιγμή λοιπόν που θα εκπνεύσει αυτή η εξαίρεση ο κανονισμός τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι σε απόλυτη εφαρμογή και θα υπάρχει καμία ανοχή για αυτή την εξαίρεση. Και τέλο, τα ποσά τα οποία δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Μαρόκο για να καταργηθούν αυτά τα παρασυρώμενα δίκτυα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν το ταχύτερο ώστε το πρόβλημα αυτό να επιληθεί επιτέλου. Αυτά είναι τα σχόλια που ήθελα να σας κάνω κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την Κομισιόν, λέει και η πρόεδρο. Θέλω να σα υπενθυμίσω ότι έχω ένα σημείωμα της γραμματείας σε σχέση με τα πορίσματα της συνεδρίασης της ΙΚΑΤ. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να κλείσουμε το σημείο αυτό της ημέρησης διάταξης και τώρα αυτό το οποίο θα αναζητήσω στον κύριο Ρωμέβα είναι σε 5 λεπτά να αντιμετωπίσει τον 13ο πρόγραμμα τεκμηρίωσης για τον ε, γαλαζόπτερο τόνο ή εδώ γιατί σε 10 λεπτά πρέπει να ξεκινήσει και η ακρόασή μας. Εγώ είχα ζητήσει κάτι πάρα πολύ απλό. Ήθελα να ξέρω από την Κομισιόν, μετά από τα συμπεράσματα της ΕΚΑΤ, ποιες ήταν οι αλλαγές οι οποίες θα επιφέρθουν. Γιατί το πρόβλημα που έχω είναι ότι στη δική μου έκδοση του κειμένου έχω απλώς ένα σχέδιο της ε, θέσης της Κομισιόν. Θα ήθελα να ξέρω αν η Κομισιόν μπορεί να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τις συγκεκριμένες αλλαγές οι οποίες προκύπτουν από τη συνεδρίαση της ΙΚΑΤ. Γιατί έχω τρία σχέδια στα χέρια μου, δεν ξέρω ποια από τα τρία είναι το οριστικό το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή. Δεν ήθελα λοιπόν να λάβω το λόγο εγώ ο ίδιος, απλώς ήθελα να ακούσω από την πλευρά της Κομισιόν και από τα χείλη της ποιες θα είναι οι αλλαγές που θα υπάρχουν. Κύριε Κέμφ, θέλετε να μας πληροφορήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος σε σχέση με τις αλλαγές στο κανονισμό για τις ε, αλλιεύματα του κόκκινου τόνου. Το θέμα είναι τεχνικό, δεν άλλαξε. Όπως είπε ο συνάδελφος, κυρίως πρόκειται για ενίσχυση ορισμένων πτυχών του συγκεκριμένου προγράμματος. Οι αλλαγές είναι η αρχή του διαχωρισμού των αλλιευμάτων. Δηλαδή τα αλλιεύματα θα πρέπει να ξεχωρίζονται ανάλογα με κράτος σημαίας αν ένα συμβαλόμενο μέρος είναι τρίτης χώρας, έπειτα είναι ο διαχωρισμός των αλλιευμάτων με βάση το έτος, δηλαδή οι διατάξεις της ΕΚΑΤ ενισχύθηκαν για να μην έχουμε αυτή την ανάμειξη, δηλαδή τα ψάρια αυτά πρέπει να θανατώνται την ίδια χρονιά στην οποία αναλιεύθηκαν ή να μην υπάρχει δυνατότητα να θανατώνται πριν το την αρχή της επομένης περίοδου αλίευσης και ορισμένες μέθοδοι δεν επιτρέπουν τη θανάτωση πριν από την αρχή της νέας περίοδου. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει μια δήλωση αναβολής των αλλιευμάτων. Δηλαδή αν σε μια συγκεκριμένη χρονιά, σε μια συγκεκριμένη μονάδα γίνεται ανάμειξη των αλλιευμάτων, η κλωβή θα πρέπει να είναι σαφώς διαχωρισμένη. Άλλο στοιχείο στο παράρτημα είναι κάτι πολύ πιο πρακτικό για την εφαρμογή του προγράμματος και αφορά την πώς συμπληρώνεται το έντυπο. Δηλαδή η βάση του προγράμματος στηρίζεται σε ένα έντυπο μετά την αλλιεύματα, από την, από την αλλίευση μέχρι την τελική εισαγωγή. Το έντυπο πρέπει να συνοδεύει τον κόκκινο τόνο. Κάθε φορέας θα πρέπει να συμπληρώνει το κομμάτι του εντύπου που τον αφορά με συγκεκριμένες οδηγίες σε παράρτημα ο καθένα λοιπόν ξέρει ποια στιγμή πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο και η κυβέρνηση ξέρει ποια στιγμή πρέπει να επικυρώσει το έντυπο. Προσθέθηκε και ένα πρακτικό τμήμα στο πρόγραμμα για ορισμένε δυσκολίες που είχαμε γιατί οι φορεί οι ίδιοι μας το ζήτησαν. Σαφή κανόνα δηλαδή. Και σύντομα να απαντήσω στα θέματα που έθεσε ο κύριος Ρωμέβα για τα κατεψυγμένα. Φυσικά το πρόγραμμα καλύπτει τα νοπά, τα κατεψημένα και τα σε υπερκατάψυξη. Μετά τη θανάτωση το προϊόν μεταφέρεται με πλοία που κάνουν την επεξεργασία στο πλοίο, οπότε η κατάψυξη γίνεται στο πλοίο. Στην περίπτωση αυτή το πρόγραμμα εφαρμόζεται και στο κατεψυγμένο προϊόν, δηλαδή το έντυπο πάνω στο πλοίο μένει μέχρι τη χώρα εισαγωγής, που συνήθως είναι η Ιαπωνία, Άρα καλύπτονται και τα κατεψυγμένα προϊόντα. Τώρα για την αποθήκευση των κατεψυγμένων προϊόντων. Πέρυσι στο Μαρακές προτείναμε να έχουμε ένα μητρό εισαγωγών με το αριθμό των αποθηκών που έχουν, ψυγεία αποθήκες. Δυστυχώς το μέτρο αυτό δεν εγκρίθηκε από την ΕΚΑΤ στο τι συνέχεια δίνεται, τι παρακολούθηση δηλαδή ως προς τα κατεψυγμένα προϊόντα, συμφωνούμε ότι επιδέχεται βελτίωση του σύστημα. Πρέπει να ξεκινήσουμε από, τον, από το Μητρό. Πάντως φέτος δεν εγκαταλείψα ακόμα την ιδέα. Ο έλεγχος στην εισαγωγή να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της ΕΚΑΤ σε μια πιο τεχνική ομάδα εργασίας ενδιάμεσα. Η ενίσχυση λοιπόν των ελέγχων στην εισαγωγή και μιλάμε κυρίως για την Ιαπωνία είναι προτεραιότητα. Θα συζητηθεί. Πάντως το θέμα των κατεψυγμένων αποθηκών και των κατεψυγμένων προϊόντων είναι και αυτά τμήμα της συζήτησης. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ρωμέβα, δεν θέλετε να κάνετε κάποια παρατήρηση. Εντάξει. Το μόνο το οποίο σας ζητώ είναι να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα, επειδή το θέμα αυτό και αυτό θα επισέλθει στη συναπόφαση και όταν έχουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα μας βοηθήσει να εργαστούμε καλύτερα. Έτσι κλείνουμε και το 13ο σημείο της ημερήσιας διάταξης και περνάμε τώρα στην ε, ακρόαση με 5 λεπτά προπορία. Σας παρακαλώ να καθίσετε όλοι. Πρόκειται για τη δημόσια ακρόαση για την πράσινη βίβλα που αφορά τη μεταρρύθμιση της κοινής αλληλευτικής πολιτικής, όπως γνωρίζετε πολύ καλά. Όλοι οι παρόντες και πάλι βρισκόμαστε ενώπιον μιας σημαντικής προκλήσεως που είναι η τροποποίηση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής και έχουμε προσκαλέσει σήμερα ένα μεγάλο μέρος από τους εκπροσώπους των αληφτικών φορέων του τομέα οι οποίοι θα μας παρουσιάσουν τις θέσεις τους και τις απόψεις τους σε σχέση με την Πράσινο Βίβλο. Φυσικά θα κάνουμε και άλλες τρεις ακροάσεις το επερχόμενο έτος σε σχέση με τα βασικά θέματα της διαχείρισης και της προστασίας για την εμποροποίηση και τα λοιπά για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις νομοθετικές προτάσεις οι οποίες θα προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Επίτροπη. Προς το παρόν εμείς είμαστε στο πλαίσιο του, της Πράσινης Βίβλου. Ξέρετε ότι η κυρία Πετράου Νέβης είναι αυτή η οποία είναι συγγήτρια από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα είμαι εξαιρετικά αμήλικτη με τους χρόνους αγόρευσης γιατί είναι πάρα πολύ καλεσμένοι μας και πολύ λίγος ο χρόνος της συνεδρίασής μας. Γι' αυτό σας ζητώ να σεβαστείτε απόλυτα το χρόνο μιλίας σας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παρόντες για την παρουσία τους σε αυτήν την ακρόαση και δίνω για πέντε μόνο λεπτά το λόγο στην κυρία Πατράου Νέβης, η οποία είναι συγγήτρια για αυτό το θέμα. Κυρία Πατράου, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω την τιμή και την ευθύνη να είμαι η για αυτό το συγκεκριμένο, για αυτό το σημαντικό θέμα που είναι η πράσινη βίβλος της Κομισιόν σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει μεταρρυθμιστής κοινή πολιτικής αλίας ενώπιον όλων των συναδέλφων μου, αλλά κυρίως ενώπιον των εκπροσώπων του αληφτικού τομέα. Είναι πραγματικά μια μεγάλη τιμή να μπορώ να λάβω το λόγο. Θέλω να χαιρετήσω όλους τους παρόντες και θέλω να σας πω ότι το έργο το οποίο θα πρέπει να φέρει σε πέραση η Επιτροπή Αλίας για το ζήτημα της Πρασίνης Βίβλου είναι ήδη πάρα πολύ εντατική εργασία μας. Είχαμε ήδη μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων τον Οκτώβριο, μια δεύτερη τον Νοέμβριο και χθε ακόμα είχαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων επί τη βάση ενός εγγράφου εργασίας το οποίο είχα την τιμή να παρουσιάσω η υποφαινομένη. Μπορώ να σας προσθέσω επίσης ότι μετά από την επεξεργασία που έχει λάβει χώρα στην Επιτροπή μας του εγγραφού αυτού μπορούμε να διακρίνουμε ορισμένους ευρύς τομείς συνένεσης για τα θέματα αυτά. Συμφωνούμε λοιπόν ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε μια τριλογία επιταγών για το μέλλον. Καταρχήν η προστασία των ε, αλλιευτικών πόρων και του περιβάλλοντος, η υποστήριξη σε κοινωνικό επίπεδο των αλλιέων <clears throat> και των εσόδων τους και φυσικά η συνολική οικονομική διάσταση της αλλιές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά τα τρία στοιχεία θα πρέπει να συγκλίνουν και να εξασφαλίσουν μια ισορροπία, μια ισορροπία που θα είναι φυσικά δυναμικού χαρακτήρα, αλλά πέραν, αν δεν υπάρξει μια τέτοια ισορροπία, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την αηφορία και την ανάπτυξη του αλληλευτικού τομέα. Θεωρώ ότι για να μπορέσουν να υλοποιηθούν αυτές οι γενικές αρχές, απαιτείται μια συγκεκριμένη <clears throat> διαδικασία αποκέντρωσης της διαχείρισης των αλλιευμάτων που σημαίνει ότι θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνε στις διάφορες περιοχές όπου λαμβάνει η χώρα η Αλία και απαιτούν την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε τις απαράγραπτε συνθήκες για μια πολιτική συμμόρφωση και υπεύθυνοποίηση που είναι αυτό το οποίο ζητούμε όλοι. Επιπλέον λοιπόν αυτών των γενικών γραμμών που ανέφερα προηγουμένως θα πρέπει να τονίσω ότι κανένας άλλος τρόπος δεν μπορεί να εξασφαλίσει την αηφορία και την διατήρηση των αλληλευτικών πόρων. Κάτι ακόμα που θέλω να προσθέσω είναι ότι πιστεύω ότι υπάρχει επίσης ευρεία συνένεση σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ότι χρειάζεται καταρχήν να υπάρξει μεγαλύτερη επένδυση για τις επιστημονικές έρευνες που θα πρέπει να αποτελέσουν το υπόβαθρο των αποφάσεων οι οποίες θα ληφθούν στον τομέα της μελλοντική ευρωπαϊκής πολιτικής αλίες. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη διατήρηση και την αηφορία των ε, αλληλευτικών πόρων, όπως είπα προηγουμένως. Θα πρέπει να υπάρξει η αποκέντρωση των διαχειριστικών μέτρων που πιστεύουμε ότι θα είναι ευεπίφοροι για μια καλύτερη πολιτική συμμόρφωση και υπευθυνοποίηση όλων των εμπλεκομένων είναι απαραίτητη επένδυση και στον έλεγχο και την εποπτεία των αλληλευτικών δραστηριοτήτων. Η μελέτη αντικτύπου επί τη βάση διαφορετικών υποδειγμάτων διαχείρισης δεν θέλουμε να διατηρήσουμε στο διηνεκές τον ηγεμονικό χαρακτήρα ενός συστήματος που βασίζεται σε συνολικά λιεύματα και ποσοστό, θέλουμε να εξετάσουμε και άλλα συστήματα τα οποία μπορεί να είναι πιο πρόσφορα για ορισμένε περιοχές και ορισμένα είδη αλίες, Επίσης, <clears throat> να προβλεφθεί η δυνατότητα διαφοροποιημένων μέτρων σε ό,τι αφορά τον βιοτεχνικό στόλο αλίας έναντι του βιομηχανικού στόλου αλίας. Επίσης, μια μεγαλύτερη προσοχή για την, ε, ε για την υδατοκαλλιέργεια, καλύτερη ανιχνευσιμότητα για τα αλλιεύματα είτε προέρχονται από την υδατοκαλλιέργεια είτε προέρχονται από την αλλία και φυσικά και μια μεγαλύτερη ενσωμάτωση της κοινή ε, οργάνωσης αλλίας στην ευρωπαϊκή πολιτική θαλασσίων πόρων. Δεν έχω φυσικά το χρόνο να σας παρουσιάσω όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά και είναι και η κατάλληλη στιγμή να ακούσουμε περισσότερο τη φωνή των εμπλεκομένων φορέων στον τομέα αλίας που είναι σήμερα προσκεκλημένοι μας και που η συμβολή σας θα είναι σίγουρα αποφασιστική για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτή την εργασία η οποία είναι ήδη πάρα πολύ εντατική με πίεση χρόνου γιατί θέλουμε μέχρι τις 11 του μηνός να ολοκληρώσουμε αυτό το έγγραφο στην Επιτροπή Αλίας. Θέλω και επανέφευχαριστήσω όλους αυτούς που είναι παρόντες στη σημερινή ακρόαση και θέλω να τονίσω και πάλι το τελείως ανοιχτό πνεύμα που έχω για να ακούσω με μεγάλη προσοχή όλες τις προτάσεις που έχετε να διατυπώσετε και θα τις συμπεριλάβω στο βαθμό του δυνατού στην έκθεση της Επιτροπής Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να βελτιώσουμε και το περιεχόμενο τους, που είναι κάτι το οποίο όλοι φυσικά πιστεύω ότι επιθυμούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πετραουνέβης. Ακολουθεί τώρα εξ ονόματος της Γενικής Διεύθυνσης ε, Αλίας, ο κύριος Φωτιάδης. Έχετε πέντε λεπτά χρόνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάνω Έχει Έχουμε ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες μας για, το πρώτο, για την πρώτη φάση της ε, μεταρρύθμισης. Έχουμε την, λευκή, την ε, πράσινη βίβλο. Μέχρι τη στιγμή που εξεδόθη η Πράσινη Βίβλος είχε οργανώσει περίπου 100 σεμινάρια Ευρωπαϊκή Ένωση με προσώπους των κρατών μελών, με φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως με τους επαγγελματίες του κλάδου για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να εμβαθύνουμε την ε, προβληματική σε σχέση με τα θέματα αυτά. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε 14 συμπληρωματικές συνεδριάσεις και θα έχουμε επομένως φτάσει στο να έχουμε ακούσει τις απόψεις όλων των κρατών μελών και όλων των εμπλεκομένων φορέων στον τομέα της αλίας και της μεταποίησης για τις προτάσεις της Κομισιόν. Στόχος μας είναι να συζητήσουμε, να αναλύσουμε όλα αυτά τα θέματα, αλλά κυρίως να μπορέσουμε να εντοπίσουμε εναλλακτικές επιλογές οι οποίες θα μπορούσαν να τύχουν επεξεργασίες στις μελέτες αντικτύπου, οι οποίες είναι εν αυτή τη στιγμή. Αυτές είναι μελέτες σε βάθος. Έχει ξεκινήσει η πρώτη, ήδη η διαδικασία. Έχουμε 30 εμπειρογνώμονες που εξετάζουν το τωρινό σενάριο, το status quo και περιμένουμε στα μέσα ε, Ιανουαρίου, αρχές Ιανουαρίου να έχουμε τα πορίσματά τους. Από το Φεβρουάριο τα πορίσματα αυτά θα γίνουν δημόσια και η Επιτροπή θα περάσει στο δεύτερο στάδιο αυτής της ε, έκθεσης αντικτύπου. Μέχρι το καλοκαίρι περίπου 40 εμπειρογνώμες θα αναλύσουν όλες τις εναλλακτικέ ε, προτάσεις, τα σενάρια τα οποία έχουν προταθεί από τα κράτη-μέλη και τους φορείς σε μια φάση διαλόγου και διερεύνησης <clears throat> όπως ελέγχθη. Η διαδικασία της Πράσινης Βίβλου είναι μια αρκετά συνολική διαδικασία. Προσπαθούμε να έχουμε μια ανάλυση η οποία θα αναλύσει όλα τα θέματα χωρίς ταμπού. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να μπορούμε να αναλύσουμε όλα τα εμπλεκόμενα προβλήματα και συμφέροντα. Η διαδικασία αυτή λοιπόν θα καταλήξει σε μια πρόταση <clears throat> από την πλευρά της Κομισιόν των συμπερασμάτων από αυτή τη φάση διαλόγου. Το πρώτο τρίμηνο του 2010 έχει προβλέψει η Κομισιόν να περατωθεί αυτή η διαδικασία και τον Απρίλιο το Συμβούλιο των Υπουργών θα διοργανώσει ένα συνέδριο Υπουργών για αυτή την προβληματική. Πιστεύουμε ότι μέσα από αυτή τη συζήτηση μπορούν να προέλθουν οι κύριοι άξονε τη μελλοντική πολιτική και αυτό θα γίνει το Μάιο όταν η Ισπανική Προεδρία έχει προβλέψει μια συνεδρίαση στην Λα Κορούνια 2 και 3 Μαΐου για τα θέματα μεταξύ των επαγγελματικών κλάδων αλίας και ένα συμβούλιο αλίας στο Βίγο την ε, επαύριο αυτή τη συνεδρίαση. Θέλουμε λοιπόν να οδηγήσουν όλα αυτά σε, ένα, σε μια λευκή βίβλο και ένα πρόγραμμα, ένα, μια πρόταση μάλλον κανονισμού που θα εκδοθούν στο τέλος του 2010, αρχές του 2011 και θα είναι η απόλυξη αυτής της συζήτησης. Μέσα στο πλαίσιο λοιπόν της τρέχουσα συνεδρίασης θέλω να σας τονίσω μόνο σαν στοιχείο συζήτηση, γιατί δεν έχουμε ακόμα λάβει οριστική θέση, ότι έχουμε εντοπίσει τέσσερα βασικά στοιχεία προβληματισμού πέρα, πέριξ των οποίων μπορούμε να αρθρώσουμε τη συζήτηση. Καταρχήν το θέμα της ευκυβερνησίας. Με ποιο τρόπο θα εξασφαλίσουμε την καλύτερη διαχείριση της λήψης απόφασης, την περιφερειοποίηση ή αποκέντρωση της λήψης απόφασης. Αυτό είναι το ένα θέμα το οποίο συζητούμε με τα κράτη-μέλη, με όλους τους εμπλεκομένους και αυτό φυσικά έχει μια κεφαλαιόδη σημασία για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία προβλέπονται στην Πράσινη Βίβλο για μια μελλοντική πολιτική η οποία να είναι πιο κοντά στον τομέα αυτό, πιο κοντά στην πραγματικότητα, την επιτόπια και που να λαμβάνει υπόψη τη διαφοροποίηση και τι ιδιαιτερότητε των περιοχών στι οποίε ασκείται η ελευτική δραστηριότητα. Αυτή η διαδικασία λοιπόν θα μα οδηγήσει σε τροποποίησει, οι οποίε θα βρίσκονται μέσα στα πλαίσια τη διαδικα... τη ε, συνθήκης της τόσο σε ό,τι αφορά την αποκέντρωση προς τα κράτη-μέλη όσο και τη μεγαλύτερη υπευθυνοποίηση του τομέα και την δυνατότητα επίσης να δημιουργηθούν περιφερειακά φόρουμ για συζήτηση και προτάσεις ακολουθώντας την, ε, <clears throat> τις ε, ρήτρε της ε, συνθήκης Λισαβόνας και σύμμορφα με τους στόχους που έχουμε θέσει στον εαυτό μας. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο έχει εντοπίσει η Κομισιόν είναι η ανάγκη να τροποποιηθούν μηχανισμοί πρόσβασης και διαχείρισης των αλληλευτικών πόρων. Προφανώς θα είναι διαφορετική λογική που αφορά την βιομηχανική αλληλεία και τη βιοτεχνική αλληλεία. Και φυσικά τίθεται επιτάπητος όλη η πολιτική επιδοτήσεων, η πολιτική χρηματοδότησης και η εξωτερική διάσταση της δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτοί οι τέσσερις άξονες είναι το κέντρο του προβληματισμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα η κυρία Σάντσεφ Τρούχη Γιάννο από την Ισπανική Προεδρία που είναι η Γενική Διευθύντρια στην Γενική Γραμματεία των Θαλασσίων Θεμάτων. Κυρία Σάντσεφ, σας δίνω το λόγο. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη ικανοποίηση για μένα να συμμετέχω σε αυτή τη συνεδρίαση τη Επιτροπή Αλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αντιμετωπίζει το θέμα τη μελλοντική πολιτική αλία. Η Ισπανία Προφανώ έχει μεγάλο ενδιαφέρον στην πολιτική αλίας και στην νέα αυτή μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική ω επερχόμενη προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε την πρόθεση να αντιμετωπίσουμε την ανάλυση όλων αυτών των θεμάτων μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2010. Προ το παρόν, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει τροποποίηση τη κοινή αλληλευτική πολιτική, διότι έχουμε νέε υποχρεώσει οι οποίε προκύπτουν <clears throat> και επειδή υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τώρα τη διαδικασία λήψη αποφάσεων καθώ και τι προοπτικέ του τομέα αυτού. Από το 2002 μέχρι το 2009 Λόγω διεθνών υποχρεώσεων ή λόγω ιδία πρωτοβουλία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει μια σειρά υποχρεώσεων που θα έχουν σαφώ αντίκτυπο στη λειτουργία τη κοινή αλληλεγγύη πολιτική και που θα αναφερθώ σε αυτού του τομεί στη συνέχεια. Καταρχήν, μια συστημική προσέγγιση, μια ολοκληρωμένη ε, αντιμετώπιση, μια αηφόρος διαχείριση, η αντιμετώπιση των απορρίψεων ηχθείων, όλα αυτά είναι τα κομβικά στοιχεία της νέας αλληλευτικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα της μείωσης των απορρίψεων όμως δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αποκλειστικό και μόνο σαν μια βελτίωση της επιλεκτικότητας των αλληλευτικών μεθόδων, γιατί πολλές φορές οι απορρίψεις οφείλονται στην έλλειψη ποσοστώσεων είτε γιατί τα κράτη-μέλη έχουν εξαντλήσει αυτές τις ποσοστώσεις, είτε γιατί δεν έχουν επαρκείς ποσοστώσεις. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια απόλυτα, απόλυτη υποχρέωση να απορριφθούν και πάλι τα ψάρια στην ε, θάλασσα, γιατί αλλιώς επικρέμανται κυρώσεις στους αλείς και στο κράτος μέλος. Ένα σύστημα αλίας λοιπόν το οποίο βασίζεται σε συνολικά αλιεύματα και ποσοστώσεις θα πρέπει να τύχη μεταρρύθμισης μέσα στα πλαίσια μιας πολιτικής πολυ... πολυεδρική σε σχέση με την αλία, δηλαδή σύλληψης πολλαπλών ειδών. Αυτό δεν μπορεί να είναι συμβατό με την τωρινή πολιτική απόρριψη των νυχθείων. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα να υπάρχουν παράλληλες μορφές αλίες, αλλά εάν δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες ποσοστώσεις για αυτές, ο κίνδυνος περαιτέρω απορρίψεων παραμένει. Είναι απαραίτητο λοιπόν να δώσουμε έμφαση στα όρια αλληλευτικής ικανότητα. Αυτό είναι ένα σύστημα το οποίο είναι πιο εύκολο να το ελέγχει κανείς βασιζόμενοι στις τωρινές συνθήκες που υπάρχουν στους αλληλευτικούς στόχους. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί πράγματι ο αλληλευτικός στόλος να δηλώνει όλα τα συλλεγόμενα αλληλευτικά είδη και θα δίνει πολύ περισσότερα στοιχεία στους επιστημονικούς φορείς για να μπορέσουν να αναλύσουν την εξέλιξη των αλληλευτικών πόρων. Ένα τέτοιο σύστημα λοιπόν που βασίζεται σε οροφές αλλιευτικής ε, ικανότητας, αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί στις περιπτώσεις μόνο κατά κάποιο τρόπο με για ένα μονάχα είδος όπου υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών που λαμβάνει η χώρα αυτή η αλία και των ειδών τα οποία αλλιεύονται. Όλες αυτές λοιπόν οι αντιμετωπίσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε μια νέα προσχέγγιση στην κοινή αλλιευτική πολιτική. Εξάλλου, η διαχείριση των διαφορετικών ειδών αλίας μπορεί να είναι και μια λύση για τις επιχειρήσεις που ασκούν την αλία γιατί μπορούν να έχουν μια μεγαλύτερη ευκαμψία σε σχέση με τον τρόπο που επενδύουν στον τομέα αυτό. Το σύστημα αυτό όμως δεν φαίνεται ότι είναι το πιο πρόσφορο για την παράκτια και βιοτεχνική αλία που είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και εκεί θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνικο-οικονομική πτυχή. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι είναι απαραίτητο η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει την απαραίτητη ε, έμφαση στην πολιτική αυτή και στην ενσωμάτωσή της στις γενικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συμφωνίες με τρίτες χώρες όχι μόνο πρέπει να συνεχιστούν αλλά θα πρέπει να ενισχυθούν επίσης. Η μεταρρύθμιση λοιπόν Τη κοινή αλληλευτική πολιτική θα πρέπει να έχει και μια εξωτερική πτυχή, μια ενίσχυση των ε, εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μα, των περιφερειακών συμφωνιών διαλύε, μια επικαιροποίηση και εδραίωση αυτών των αρχών που πρέπει να διέπουν αυτέ τι συμφωνίε τη υπεύθυνη αλληλεία και επίση τη διατήρηση σε διεθνέ επίπεδο του Ευρωπαϊκού Αλληλευτικού Στόλου. Όπως ξέρετε, θα αναλάβει τη σκητάλη η Ισπανική Προεδρία. Προβλέπεται στα συμβούλια του Απριλίου και του Ιουνίου να αντιμετωπιστεί το θέμα της μεταρρύθμισης κοινή αλληλευτικής πολιτικής που θα συμπληρωθεί με αυτή την τομεακή συνδιάσκεψη που θα γίνει το Μάιο, της οποίας θα ακολουθήσει το Συμβούλιο Υπουργών του Μαΐου. Θέλω επίσης να σας τονίσω ότι όπως γνωρίζετε έχει προβλεφθεί να είναι μια αντιμετώπιση κατά τρόικες προεδριών η Ισπανία, το Βέλγιο και η Ουγγαρία, λοιπόν, τρει επερχόμενε προεδρίε θα έχουν στο κέντρο των προσπαθειών του για την αλία ακριβώ αυτή τη μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και σα ευχαριστούμε που σεβαστήκατε και το χρόνο αγόρευση. Δίνουμε τώρα το λόγο στου προ και κλειμένου μα με την εξή σειρά. 10 λεπτά στον κύριο Παστόρ, ο οποίο είναι ο πρόεδρο τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Αλία και την Κατοκαλλιέργεια και της ε, Ένωσης για την μεταποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δέκα λεπτά. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στα δέκα λεπτά που έχω θα προσπαθήσω να, μετα... να σας μεταδώσω την αίσθηση που έχει αναπτύξει η ΕΚΦΑ ε, σχετικά με τις προτάσεις ε, της Κομισιόν. Δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες όπως καταλαβαίνετε. Νομίζω όμως ότι μπορώ να εκφράσω κάποιες βασικές κατευθύνσεις συλλογισμού. Να σας θυμίσω καταρχήν ότι η ΑΚΦΑ είναι ένα φόρουμ που αποτελείται από πολλούς διαφορετικούς φορείς. Ε, δεν πρόκειται λοιπόν μόνο για τους οικονομικούς φορείς. Ε, εκπροσωπούνται και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Δημιουργήσαμε μια ομάδα εργασίας ειδικά για να εξετάσει τις προτάσεις αυτές. Είχαμε αρκετές συναντήσεις φέτος για να εκπονήσουμε ένα έγγραφο θέσης. Αυτό δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα. Μιλώ Λοιπόν, με βάση τι συζητήσει που έχουν γίνει μέχρι τώρα, η Ολομέλεια τη ΑΚΦΑ την επόμενη εβδομάδα ελπίζουμε θα μπορέσει να υιοθετήσει την έκθεση αυτή και να την λάβετε. Να λάβετε την οριστική έκθεση. Να αναφερθώ στα σημεία που θα συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση. Καταρχήν η ΑΚΦΑ συμφωνεί με την ανάλυση της Κομισιόν. Πράγματι, τα σημεία που ανέφερε είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στην αλληλευτική πολιτική αυτή τη στιγμή. Ταυτόχρονα, η ΑΚΦΑ θέλει να τονίσει ότι έχουν γίνει σημαντικέ τροποποίησει τα τελευταία χρόνια. Πολλά πράγματα έχουν γίνει όσον αφορά την αλληλευτική ικανότητα, την διαχείριση και την κατάσταση των αλληλευτικών πόρων. Η κατάσταση λοιπόν είναι αρκετά ζωφερή, υπάρχουν ε, όμως ε, και κάποια ε, σημεία που θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω. Υπάρχει μια αίσθηση ότι δεν χρειαζόμαστε πάντα νέα πολιτική, αλλά καλύτερη επιβολή της πολιτικής. Αυτά όσον αφορά το επίπεδο φιλοδοξίας μας. Ένα από τα κεντρικά σημεία στο, στη διαχείριση της αλληλείας, ε, την η ιδιοκτησία των δικαιωμάτων αλληλείας, υπάρχουν διστάμενες απόψεις σχετικά με τα βιβάσιμα δικαιώματα. Ιδιαίτερα από την αλληλεία μικρής κλίμακας, από το τομέα του αλληλεία, της αλληλείας μικρής κλίμακας υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το θέμα αυτό. Ε, κάτι τέτοιο ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει αποκεντρωμένη προσέγγιση. Θέλουμε ε, τριπλή αηφορία, ε, οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική. Εάν δεν υπάρχουν ψάρια, δεν θα υπάρχει ούτε οικονομία, ούτε ε, κοινωνική αηφορία. Θα χρειαστεί λοιπόν να θέσουμε προτεραιότητες. Θα πρέπει όμως να εξετάσουμε τις τρεις αυτές πτυχές με το σωστό τρόπο. Χρειαζόμαστε δείκτες και στόχους για την εφαρμογή των διαφόρων αυτών στοιχείων. Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να εκπονηθούν με επιστημονική βάση κατόπιν διαβούλευσης με όλους τους ενδιαφερομένους. Όπως σας είπα, η ΑΚΦΑ συμφωνεί με την αποκεντρωμένη προσέγγιση και πιστεύουμε ότι υπάρχουν δύο βασικά επίπεδα, τα ΡΑΚ, τα Περιφερειακά Συμβούλια, υπό τη που έχουμε σήμερα. Πιστεύουμε όμως ότι στο μέλλον τα ΡΑΚ αυτά θα χρειαστούν και κάποια υποστήριξη, θα χρειαστούν επιστήμονες και ανθρώπους από τις εθνικές κυβερνήσεις ώστε τα ΡΑΚ να είναι σε θέση να δώσουν πιο δεσμευτικές συμβουλές. Όσον αφορά τις ε, συμβουλές σε, ε, σε μάκρος χρόνου, οι ΡΑΚ είναι σε πολύ καλή θέση να παρέχουν ε, τέτοιες συμβουλές. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προσέξουμε να μην προσθέσουμε επίπεδο ανάμεσα στην ΑΚΦΑ και στα ΡΑΚ και να μην αυξήσουμε τη γραφειοκρατία. Η ΑΚΦΑ δεν πιστεύει ότι ο τομέας αυτός θα πρέπει να αποκτήσει περισσότερη ευθύνη μέσα από αυξημένη αυτοδιαχείριση. Όσον αφορά την αλία μικρή κλίμακα, ε, μόλι ανέφερα ότι θεωρούμε ότι είναι πολύ, πολύ ο τομέα αυτός και στις συζητήσεις μας προτείνουμε να εξεταστεί η πιθανότητα μιας πιο αναλυτικής μελέτης, διότι αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε πώς αυτό μπορεί να ταιριάξει με το σύστημα διακυβέρνησης. Υπάρχει λοιπόν εδώ σαφώς ανάγκη για περαιτέρω δράση όσον αφορά την διαχείριση της αλληλείας από την βιολογική πλευρά. Σίγουρα η ιδέα αυτή που έχει παρουσιαστεί είναι η κατάλληλη για το μέλλον. Πιστεύουμε όμως και πάλι ότι χρειάζεται περαιτέρω έρευνα για να δούμε πώς μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα ε, επίπεδα φιλοδοξίας μας είναι ρεαλιστικά, αυτά είναι, αυτό είναι σημαντικό ερώτημα για την ΑΚΦΑ. Πολύ σημαντικό θέμα είναι η μείωση των απορρίψεων, η οποία θα βελτιώσει και την εικόνα της κοινή ελληνικής πολιτικής. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όμως ε, με ένα ε, σφαιρικό πρόγραμμα διαχείρισης, θα πρέπει να ε, γίνει λεπτομερής ανάλυση. Η εκφόρτωση όλων των ψαριών ε, με υψηλότερες ποσοστώσεις ε, έχει βρει υποστήριξη. Μπορεί να μην είναι κατάλληλο αυτό για όλα τα είδη ψαριών. Πιστεύουμε, η ΑΚΦΑ όμως πιστεύει ότι μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το σύστημα σε κάποιες περιπτώσεις αλλιευμάτων. Και όσον αφορά τις ποσοστώσεις ε, θέλουμε μεγαλύτερη ευελιξία, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανταλλαγή ποσοστώσεων ανάμεσα στα κράτη-μέλη και ακόμα περισσότερο ανάμεσα στα ε, κράτη-μέλη και τρίτες χώρες ε, που αλλιεύουν στα ίδια ύδατα. Λοιπόν, η ανταλλαγή ε, ποσοστώσεων δεν έχει συζητηθεί εις βάθος. Θέλουμε όμως να εξετάσουμε τη δυνατότητα περαιτέρω ευελιξίας. Όσον αφορά την αγορά, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ εκπώνησε μία μελέτη που ολοκληρώθηκε την, τον Μάιο από την εταιρεία Ernst Young που εξέτασε την κατάσταση στην αγορά. Τέσσερις βασικές προκλήσεις εντοπίστηκαν και πιστεύουμε ότι είναι πολύ επίκαιρα τα ζητήματα αυτά. Καταρχήν, θα πρέπει να υπάρξει ε, ισορροπημένη τροφοδοσία της ε, αγοράς, ε, να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα, να τρίτον να προστατευτούν τα συμφέροντα των Ευρωπαίων καταναλωτών και τέταρτον να βελτιώσουμε τη γνώση για την αλία και τη γεωργία. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ κέρια τα ζητήματα αυτά. Και θα δείτε ότι σαν λύσεις μας είναι απαραίτητο να έχουμε μια όσο γίνεται ευρεία προσέγγιση. Αυτή τη στιγμή ε, δεν κοιτάμε την αγορά στο σύνολό της. Ε, θα πρέπει να εξετάσουμε την αγορά, να ε, αποκρινόμαστε στα μηνύματα της αγοράς και να μην ξεχνάμε ότι η ευρωπαϊκή αγορά αποτελεί μέρος της παγκόσμιας αγοράς. Ε, είναι λοιπόν ε, πολύ σημαντικό το θέμα της αγοράς. Υπάρχει και, ε, υπάρχουν και οι κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες για την απασχόληση όχι μόνο στη θάλασσα αλλά και στη στεριά. Εάν δεν τροφοδοτούνται οι σχετικές βιομηχανίες, αυτό σημαίνει ότι πολλοί εργαζόμενοι, 130.000 υπάλληλοι στη στεριά, μπορεί ε, να ε, δουν ότι κινδυνεύει ε, η θέση τους, η δουλειά τους. η τροφοδοσία των βιομηχανιών αυτών γίνεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τρίτες χώρες. Κάποιες από αυτέ τι βιομηχανίε μεταποίησης δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν εάν δεν έχουν πρόσβαση στα σχετικά προϊόντα. Επίση, όταν εξετάζουμε την αγορά, είναι απαραίτητο όχι μόνο να κοιτάμε τι τιμέ, αλλά και το κόστο παραγωγή. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τα, η αλληλεία και τα προϊόντα ε, υδατοκαλλιέργειας πρέπει να ανταγωνίζονται με άλλα ε, προϊόντα που περιέχουν πρωτεΐνη και με άλλου τομεί αγορά. Γι' αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούμε όχι μόνο στι τιμέ, αλλά και στο κόστο. Για παράδειγμα, ε, κάποιες, ε, κάποια μέτρα μπορούν να αυξήσουν το κόστος παραγωγής. Και τέλος, κυρία Πρόεδρε, η τελευταία μου παρατήρηση. Για να έχουμε αηφόρο παραγωγή στην Ευρώπη και κοιτώντας όλα τα μέτρα που λαμβάνουμε, θέλουμε να διατηρήσουμε την EFF. Η ΑΚΦΑ θεωρεί ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την πιστοποίηση τρίτων μερών και να προτείνουμε ένα σαφές ε, πλαίσιο ε, ελαχίστων προτύπων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Παστόρ. Πέντε λεπτά εδώ, Βιέν Γαράτ, πρόεδρος της Europes. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω ως πρόεδρος του EuroPES και όχι εκ μέρους της Ισπανικής Οργάνωσης που εκπροσωπώ. Έχω μια συγκεκριμένη θέση με την ΚΟΣΤΖΕΚΑ και μοιράσαμε τη δουλειά. Εγώ θα μιλήσω για ορισμένα θέματα και ο συνάδελφός μου θα μιλήσει για τα υπόλοιπα. Σε πέντε λεπτά πρέπει να μιλήσουμε τηλεγραφικά. Θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα σημεία. Πρώτον, πρόκειται για μια πολιτική που βασίζεται στις γνώσεις για την Κόζικα αυτό είναι σημαντικό θέμα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως κάναμε ως τώρα, διότι το είπε και η Κομισιόν. Δεν μπορούμε να έχουμε γνώσεις για το σύνολο των αποθεμάτων. Χρειαζόμαστε μια νομική ασφάλεια, δεν μπορούμε να συνεχίζουμε με τα τάκ, με γενικευμένες θέσεις. Χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους ανθρώπινους και οικονομικούς για να εφαρμοστεί η έρευνα. Επίσης χρειάζεται μεγαλύτερο συντονισμό των ερευνητικών προγραμμάτων. Γι' αυτό προτείνουμε να υπάρξει μια, ένας ευρωπαϊκός οργανισμός έρευνας που να τη συντονίζει αυτά. Θεωρούμε ότι η συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων είναι απολύτως αναγκαία. Άλλο θέμα, η διαχείριση των αλλιευτικών μονάδων. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μακρό πρόθεσμο πρόγραμμα διαχείρισης που στηρίζεται σε συγκεκριμένες επιστημονικές θέσεις. Θεωρούμε όμως ότι θα πρέπει να δείχνουμε ευελιξία, να δούμε ποιες είναι οι κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες ορισμένων μέτρων εσωτερικά συζητάμε το θέμα διαχείρισης της αλληλείας με βάση τα αλληλευτικά δικαιώματα. Και όπως είδαμε σε επίπεδο της ΑΓΦΑ υπάρχει σύγκληση απόψεων για τον στόλο ανοιχτή θάλασσης και τα λιμάνια, ιδιαίτερα για τον βιοτεχνικό στόλο στη Μεσόγειο, χρειάζονται εξαιρέσεις σε ορισμένα σημεία. υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ οργανώσεων των διαφόρων κρατών μελών σε ορισμένα θέματα. Υπάρχει όμως συνένεση όσον αφορά την ανάγκη μια μελέτης για τα ΤΑΚ και τις ποσοστώσει της Ένωσης. Και η μεταρρύθμιση μας δίνει μια μοναδική ευκαιρία να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα σημαντικά ερωτήματα. Γενικά είμαστε υπέρ μια maximum μείωση προοδευτικά των απορρίψεων κατά αλλιευτική μονάδα με πιλωτικά προγράμματα. Η σχετική σταθερότητα. Οι Ισπανοί κινούνται μόνοι τους και οι Ευρωπαίες και οι Κοζεκά θεωρούμε ότι δεν πρέπει να κρατηθεί αυτή η σχετική σταθερότητα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το σύστημα αυτό δεν είναι τέλειο. Αλλά αντί να καταργήσουμε το σύστημα αυτό της σχετικής σταθερότητας, καλύτερα θα είναι να έχουμε ένα πιο ευέλικτο σύστημα με μηχανισμούς ανταλλαγής των ποσοστώσεων ετήσια μεταξύ φορέων περισσότερων κρατών της Ένωσης για να ευνοηθεί η πλήρης χρήση όλων των τάκ και ποσοστώσεων. Λεβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που έγιναν στα κριτήρια τελευταία 25 χρόνια. Και το 12.000. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τον ορισμό της βιοτεχνικής παράκτιας αλίας. Θα σας μιλήσουν οι συνάδελφοι γι' αυτό μετά. Διαρθρωτική πολιτική, το μελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλίας θα πρέπει να λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία της ΚΑΛΠ. Να δούμε παραδείγματος την υποστήριξη των επιστημόνων. Τα μέτρα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καινοτομίες, επιλεκτικές μορφές αλίας, χρήση των α, απορριφθέντων ηχθείων, καλύτερες επενδύσεις με δύο λόγια. Έπειτα, τι κονδύλια χρειάζονται για να δοθεί συνέχεια στις ανάγκες της μελλοντική κοινή αλληλευτικής πολιτικής, πιλωτικά προγράμματα, περιφερειοποίηση, χρειάζεται και γι' αυτό οικονομική ενίσχυση. Δεν θα μιλήσω για την εξωτερική διάσταση ούτε για το εμπόριο, θα το κάνουν οι συνάδελφοι μετά. Ευχαριστώ πολύ. Στη συνέχεια, πέντε λεπτά, κύριος Μπρον. Grazie, grazie Presidente. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω με συγκεκριμένα σημεία στο κοινό κείμενο της Ευρωπαίας και Κοζεκά για τις διαρθρωτικές αλλαγές της πράσινης βίβλου, ιδιαίτερα για το υπερβάλλον δυναμικό. Πρέπει να μελετηθεί η διαφορετική κατάσταση στην κάθε χώρα. Δεν υπάρχει μία λύση. Γιατί κάθε χώρα έχει το δικό της στόλο, τους δικούς της πόρους η λύση νομοθετικά σε επίπεδο ένωσης για το, οικονομικό, το δυναμικό είναι σωστή. Αλλά πρέπει να γίνει μια μελέτη επικαιροποιημένη, να δούμε και άλλα κριτήρια πέρα από τα απλό κριτήριο των, του τονάζ. Άλλο σημείο είναι το θέμα των ε, μεταφερόμενων δικαιωμάτων. Όπως είπε και ο Σνάφος Παστόρ, υπάρχουν διαφορετικές θέσεις. Η μικρή αλία θεωρεί ότι ο μηχανισμός αυτός είναι επικίνδυνος ότι μπορεί να οδηγήσει σε συγκεντρώσεις των αλληλευτικών δικαιωμάτων στα χέρια λίγων επιχειρήσεων ισχυρών. Για τη βιομηχανική αλληλεία μπορεί να είναι καλό σύστημα διακυβέρνησης, αλλά όλοι συμφωνούμε ότι την επιλογή πρέπει να την κάνει η κάθε χώρα μέλος και όπου εγκριθεί πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα προστασίας. Στρατηγική στόχη η πράσινη βίβλος μιλάει για η ιεράρχηση του στοιχείου της βιολογικής διατηρησιμότητας παράγγελα με το οικονομικό και κοινωνικό σκέλος σε ίσες, ίση προτεραιότητα. Αλλά στη μεταρρύθμιση του 2002 και στην πράσινη βίβλιο λείπουν ορισμένα στοιχεία. Όσον αφορά την απασχόληση υπάρχουν αντιτιθέμενες θέσεις σε διάφορα κείμενα της Κομισιόν. Για μας η απασχόληση είναι προτεραιότητα και για την ένταξη των νέων και για τη διατήρηση της απασχόλησης με προγράμματα κατάρτισης σχεδί. Το πλαίσιο των αποφάσεων. Οι Ευρωπαίες και Κοζικά είναι υπέρ ενός συστήματος όπου το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να εγκρίνουν γενικές αρχές προσανατολισμού και κανονισμούς πλαίσιο, ενώ τις διαχειριστικές αρμοδιότητες ως προς τις προτάσεις της Κομισιόν αυτό να τις εφαρμόζουν οργανισμοί αποκεντρωμένοι κατά περιοχή ή κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας. Η μεταρρύθμιση να μην ξαναεπικεντρωθεί να επικεντρώσει μάλλον την δυνατότητα λήψη αποφάσεων μόνο στην Κομισιόν ο συμβουλευτικό ρόλος. Οι γνωμοδοτήσεις της συμβουλευτική Επιτροπής Αλίας θέλουμε τακτικά να λαμβάνουν υπόψη, ακόμα και αν πρόκειται για αρνητική απάντηση. Να υπάρχει μία απάντηση πάντα. Η Συμβουλευτική Επιτροπή είναι το μόνο τυπικό όργανο διαβούλευσης για την Ένωση και παραξενευόμαστε για το ότι δεν γίνεται καν ο παραμικός υπενιγμός στην Πράσινη Βίβλο στον κοινωνικό διάλογο. Η Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου πρέπει να ζητείται η γνώμη της όσον αφορά τη μεγαλύτερη ευθύνη των φορέων υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στο σύστημα, σύστημα bottom-up της Πράσινης Βίβλου και το σύστημα ελέγχου και διαχείρισης στον οποίο αναφέρεται ο πρόσφατος κανονισμός ελέγχου, όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο. Εμείς δεν είμαστε υπέρ της πληρωμής των δικαιωμάτων αλλίας. Ήδη υπάρχει κόστος γι' αυτό, ιδιαίτερα όσον αφορά τον έλεγχο. Όλοι ξέρουμε ότι ζούμε μια κρίση, η κοινή αλλιευτική πολιτική πάει προς την κατάργηση των ενισχύσεων, συζητούνται συμφωνίες εταιρικής σχέσης, οπότε δεν μπορούμε να βάλουμε επιπλέον βάρη στα δικαιώματα αλίας. Για τη μικρή αλία τώρα πρέπει να προστατεύεται και λόγω της κοινωνικο-οικονομικής και πολιτιστικής αξίας που έχει ιδιαίτερα στη Μεσόγειο. Πρέπει πρώτα-πρώτα να γίνεται μια αξιολόγηση κοινωνικο-οικονομική. Τέλος για το διαφοροποιημένο καθεστώς δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε διαφοροποιημένη βάση κατά περιοχή. Προσοχή λοιπόν στην μικρή παράκτια αλία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πολύ προσοχή στις επιλογές που έχουμε. Τα λέμε αυτά στο κείμενό μας. Προσοχή στον αρνητικό ρόλο της ε, αθλητικής αλίας, όπως θα την έλεγα, σε σχέση με την μικρή συστηματική αλία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Μπομφίλιο. Πέντε λεπτά Φιλίπ Αλφόνσο, γραμματέας της ETF Transport Workers Federation. Πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε τη δυνατότητα να λάβουμε το λόγο ενώπιόν σας. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω το ρόλο της συνομοσπονδίας μας. Είμαστε μια πανευρωπαϊκή ομοσπονδία στον τομέα των μεταφορών και της αλίας. 2,5 εκατομμύρια εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη εκπροσωπούμε από πάνω από 200 συνδικάτα που ενεργοποιούνται σε πάνω από 40 χρόνια. Είμαστε μια λοιπόν τομεακή ομοσπονδία μέσα στην Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδεκάτων και υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των εργαζομένων στις μεταφορές και των εργαζομένων επίσης στην αλία και παίζουμε και ένα σημαντικό ρόλο για την ε, επαφή αυτών των εργαζομένων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να θεωρήσετε ότι εγώ δεν έχω ιδιαίτερη εστίαση σε αυτά που θα πω στην πράσινη βίβλο της Κομισιόν. Αυτά τα οποία θέλω να πω σήμερα μπορεί να σας φανούν λιγάκι εκτός πλαισίου. Αλλά έχω την ευκαιρία να σας μιλήσω για ένα σημαντικό στοιχείο, για να ελείποντα κρίκο στην πράσινη βίβλο που νομίζω ότι πρέπει παρόλα αυτά να ληφθεί υπόψη, που είναι η κοινωνική διάσταση τη ε, ευρωπαϊκή πολιτική αλλία. Η μεταρρύθμιση του 2002 ήταν μια χαμένη ευκαιρία για να μπορέσει η ευρωπαϊκή πολιτική αλλία να έχει μια πραγματική κοινωνική διάσταση. Σήμερα έχουμε την πρόσκληση να αντιμετωπίσουμε την αηφορία αυτή τη πολιτική. Η πράσινη βίβλο ορισμένε φορέ παρακάμπτει θέματα που είναι τόσο σημαντικά όσο η επαγγελματική κατάρτιση, τα επαγγελματικά προσόντα, συνθήκες ζωής και εργασίας πάνω στα σκάφη, τα λευτικά, θέματα υγείας και ασφάλειας, η ελκυστικότητα του τομέα αυτού και η δυνατότητά του να προσελκύει και να διατηρεί εργαζομένους στον αλληλευτικό τομέα, νομίζω ότι όλα αυτά παίζουν κάποιο σημαντικό ρόλο και η αλληλευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να τονίσουμε ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί εξ αρχής σε μια πολιτική που λαμβάνει υπόψη την κοινωνική πτυχή. Περισσότερο μια τεχνοκρατική, διαχειριστική πολιτική σε σχέση με τους αλληλευτικούς πόρους και την αλληλευτική προσπάθεια έχει αντιμετωπιστεί και μια αλληλευτική πολιτική. Νομίζω ότι η επικείμενη μεταρρύθμιση είναι λοιπόν μια ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε από πολύ κοντά όλη την κοινωνική προβληματική. Η πράσινη βίβλος δεν αντιμετωπίζει δεν παρακάμπτει απόλυτα το πρόβλημα αυτό, αλλά δεν το αντιμετωπίζει επαρκώ. Για μα τα κλειδιά μια πραγματική αντιμετώπιση κοινωνική διάσταση είναι η ενίσχυση τη επαγγελματική κατάρτιση, η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, περισσότερη βοήθεια για την ε, α, αναπροσαρμογή των ε, αλλιευτικών περιοχών. Οι προσπάθειε που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι άτολμες και περιορισμένες. Πρέπει να δοθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση και να ληφθεί υπόψη σε συνολικό επίπεδο η κατάρτιση για τα θαλάσσια επαγγέλματα. Έχουμε διαπιστώσει ότι σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο υπάρχει όλο και μεγαλύτερη προσφυγή σε μεταναστεύοντες εργαζόμενους και δεν έχουμε πρόβλημα όσο αυτό περιλαμβάνεται σε πραγματικές συλλογικέ συμφωνίες και κοινωνικό διάλογο, αλλά θα πρέπει να ληφθούν όλα υπόψη για να αποφύγουμε να καταλήξουμε σε μια πολιτική κοινωνικού ντάμπινγκ. Πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο και για τον τρόπο με τον οποίο θα υπάρξει εξυγχρονισμό του αληφτικού στόλου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπάρχει μεγαλύτερη κατάρτιση, να δημιουργηθούν οι διάβλοι που είναι απαραίτητοι μεταξύ των διαφόρων επαγγελμάτων στου ε, θαλάσσιου τομεί και να εξασφαλίσουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την τεχνογνωσία που έχουν οι εργαζόμενοι στη θάλασσα. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να υπογραμμίσω επίση είναι η ανάγκη να αναπτύξουμε μια πραγματική κουλτούρα ασφάλειας στη θάλασσα και επίσης προστασίας της υγείας. Έχουμε πολλέ φορέ πεπαλαιωμένους αλλιευτικού στόλου και είναι απαραίτητο να συλλέξουμε στατιστικά στοιχεία και να εναρμονίσουμε τις πληροφορίες που έχουμε για τα θαλάσσια ατυχήματα, να καταλάβουμε ποιε είναι οι αιτίε αυτών των ατυχημάτων. Όλα αυτά λοιπόν για μένα είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε καλύτερα τις ε, κανονιστικές ρήτρες οι οποίες έχουν εγκριθεί στην πραγματική κατάσταση των αλλιευτικών στόλων. Πρέπει επίσης να υπάρξει ενθάρρυνση στα κράτη μας να επικυρώσουν τη συνθήκη STCW και να υπάρξουν ιδιαίτερες ε, προδιαγραφές για τα σκάφη μικρότερα από 15 μέτρα μήκους. Πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν πώς θα πρέπει να διαρθρωθεί η εργασία και η αμοιβή των εργαζομένων. Υπάρχουν ε, συστήματα τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν για να εξασφαλιστούν τα έσοδα των εργαζομένων στον τομέα αυτό και επανέρχομαι στον κοινωνικό διάλογο, ο οποίο είναι κεφαλαιόδη, θα πρέπει να βελτιωθεί ιδιαίτερα, ιδίω σε μερικέ χώρε όπου είναι ανεμικός ή ανύπαρκτος ο κοινωνικός διάλογος και αυτό δεν αφορά μόνο τις πτυχές της αμοιβή των εργαζομένων αλλά και το θέμα της κατανομής των δημοσίων ενισχύσεων και των ελευτικών ε, δικαιωμάτων. Βέβαια σε πέντε λεπτά δεν μπορώ να εξαντλήσω αυτή την προβληματική όπως καταλαβαίνετε. Το ξέρω. Γι' αυτό είπαμε ότι κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους θα έχουμε σε θεματικό επίπεδο ακροάσεις για όλα αυτά τα θέματα. Μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων πάντα είναι σημαντική και νομίζω ότι ήσασταν πολύ καλός και συνοψίσατε πολύ καλά τα θέματα που θέλετε να δείξετε. Περνάμε τώρα στους προσκεκλημένους από τα περιφερειακά συμβουλευτικά ε, συμβούλια. Πρώτα απ' όλα δίνω το λόγο από το Περιφερειακό Συμβούλιο της ε, Βόρειας Θάλασσας ο κύριος Άντερσον για 8 λεπτά. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε εδώ στην Επιτροπή. Είμαι ο πρώτος ε, σε μια σειρά ε, πτά προέδρων ε, των ΡΑΚ. Ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ σήμερα είναι η μορφή της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Έχουμε αποκτήσει πείρα με τις εργασίες σε περιφερειακό επίπεδο Πάνω από πέντε χρόνια πριν ξεκινήσαμε τη δουλειά μας εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Βόρειας Θάλασσας. Και πιστεύουμε ότι έχουμε συμβάλει στην ε, βελτίωση της αλλιευτικής πολιτικής ε, τα χρόνια αυτά. Η μεταρρύθμιση της αλλιευτικής πολιτικής ε, είναι μεγάλο έργο. Δεν είναι δυνατόν σε τόσο σύντομο χρόνο να θίξουμε όλα τα ζητήματα. Θα επιλέξω λοιπόν κάποια θέματα τα οποία τίθενται προ συζήτηση. Να διαπιστώσω επίσης ότι φυσικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την μεταρρύθμιση αυτή και το δείχνει αυτό το ότι πριν ένα μήνα περίπου κάναμε μια διάσκεψη, οργανώσαμε μια διάσκεψη κατά την οποία συζητήσαμε ένα μέρος της ε, διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ε, μελλοντική αλληλευτική πολιτική. Υπήρχε μεγάλο ε, ενδιαφέρον από τους 20 εκπροσώπους που εκπροσωπούσαν όλους τους τομείς των ενδιαφερομένων στην αλληλεία. Δύο μέρες συμμετείχαν για να συζητήσουμε ακριβώς το θέμα αυτό. Δεν θα σας εκπλήξει αν πω ότι η περιφερειακή διάσκεψη της ε, αλληλευτικής πολιτικής είναι πολύ ενδιαφέρουσα για τα περιφερειακά ε, συμβούλια, τα ΡΑΚ. Με την πείρα που έχουμε αποκτήσει, μετά από πέντε χρόνια εργασία στη δική μας περίπτωση, αναπτύσσει την δουλειά που πραγματοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε με την μικροδιαχείριση, το micromanagement σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάλλον συγγνώμη ότι αυτή η μικροδιαχείριση δεν είναι βιώσιμο πρότυπο και αποτελεί έναν από τους λόγους που η παρούσα αλλιευτική πολιτική δεν έχει καταφέρει να φτάσει τους στόχους της. Αν κατάλαβα σωστά, από σήμερα εσείς εδώ στο Κοινοβούλιο συμμετέχετε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στη διαδικασία αυτή από ό,τι στο παρελθόν. Δεν πιστεύω ότι θέλετε να κάθεστε εδώ να συζητάτε μικρές μικρές λεπτομέρειες ε, σχετικά με την άσκηση της αλίας σε όλη την Ευρώπη. Στο επίπεδο αυτό θα πρέπει να συζητώνται γενικά θέματα πολιτικής. Κατόπιν θα πρέπει να ανατίθεται η διαχείριση της αλλιευτικής πολιτικής σε άλλα επίπεδα. Συνοψίζοντα την ε, διάσκεψη, μπορώ να πω ότι υπήρχε συμφωνία ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε την ε, κατεύθυνση αυτή. Υπάρχουν όμω διαφορετικέ απόψει ε, σχετικά με τα πιθανά πρότυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχουν διαφορετικέ απόψει σχετικά με το ρόλο των περιφερειακών συμβουλίων ε, στην αλλιευτική πολιτική. Μπορούμε όμω να συνεχίσουμε να το συζητάμε αυτό. Σημαντικό είναι ότι συμφωνούμε σχετικά με την κατεύθυνση της αλλιευτικής πολιτικής. είναι σημαντικό να προστατεύσουμε το πρότυπο που υπάρχει, το μοντέλο που υπάρχει. Έχουμε σε περιφερειακό επίπεδο έναν φορέα που είναι ανοιχτός για όλους τους ενδιαφερομένους. Είναι προαιρετική η συμμετοχή, είναι όμως και δυνατή η συμμετοχή για όλους. Έχουμε λοιπόν ένα διαφανές μοντέλο για να συζητάμε την βελτίωση της αλλιευτικής πολιτικής. Το 2002 ελήφθη η σχετική απόφαση και νομίζω ότι εξακολουθεί να είναι σημαντική η δουλειά των ΡΑΚ. Σημαντικό είναι να πρικοδοτηθούν σωστά τα ΡΑΚ ώστε να μπορούν να πληρούν τα καθήκοντά τους και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. Έχουμε πολύ, λίγους, πολύ ε, πενιχρούς οικονομικούς πόρους. Η διαχείριση των ε, οικονομικών θεμάτων είναι πολύπλοκη και ε, παίρνει πολύ χρόνο για μας. Νομίζω ότι μπορεί να λυθεί το ζήτημα αυτό αρκεί να υπάρχει η σχετική βούληση. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τα μοντέλα που θα πρέπει να υιοθετηθούν. Ε, θέλουμε ε, εκπροσώπηση των κρατών μελών, θέλουμε απλά ένα ε, περιφερειακό φορέα. Θέλουμε διαχείριση της αγοράς με τη συμμετοχή διαφόρων ενδιαφερομένων των κρατών μελών και της Κομισιόν. Το συμπέρασμα μου λοιπόν είναι ότι στη διάσκεψη αυτή πολλοί μίλησαν για δύο φορείς σε περιφερειακό επίπεδο. Τα ΡΑΚ δηλαδή με ενισχυμένες ε, αρμοδιότητες ε, αλλά και ε, έναν νέο φορέα. Μπορεί λοιπόν να δοθεί περισσότερη αρμοδιότητα στα ΡΑΚ. Η αυξημένη να δοθεί ε, περισσότερη ευθύνη και στη διαχείριση και στην καθημερινή αλληλεία. Στα αγγλικά υπάρχει ο όρος cultural compliance ε, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτό, να υπάρχει δηλαδή μία σειρά κανόνων ε, για την πραγματοποίηση, την εφαρμογή της αλληλευτικής πολιτικής. Κυρία Πρόεδρε, θα κλείσω σύντομα διαπιστώνοντας ότι θα συνεχίσουμε τις ε, εργασίες μας, θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στο δικό μας ΡΑΚ ε, στην ε, αλλιευτική πολιτική. Στις συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας εδώ στις Βρυξέλλες Ιταλού, όπου θα συζητήσουμε την συμβολή μας στην νέα αλλιευτική πολιτική. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε και να συζητήσουμε πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε μακροπρόθεσμες λύσεις για την αλλιευτική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Άντερσον. Στη συνέχεια, ο κύριος Γιώχανσεν, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΡΑΚ της Βαλτικής για 8 λεπτά. Ε, ε, Κύριε Πρόεδρε, κύριοι Από το 2002 ξεκίνησε ένα σημαντικό ε, πείραμα σχετικά με τη δημιουργία των ΡΑΚ. Θα ήθελα να πω εδώ στο Κοινοβούλιο ότι στην αρχή θεωρήθηκε ότι επρόκειτο για τρόπο της Κομισιόν να γλιτώσει από τα ε, σημαντικά προβλήματα και την ε, άσκηση πίεσης στους διαδρόμους από διάφορες οργανώσεις. Ε, αργότερα όμως κατάλαβε ότι δεν ισχύει αυτό. Δεν έχω πολύ χρόνο, θα προσπαθήσω όμως να διατηρήσω μια κατεύθυνση στην ομιλία μου. Είναι πολύ καλό αυτό που ξεκίνησε, αλλά στη συνέχεια δεν ε, θεωρώ ότι μπορεί να ε, συνεχιστεί αυτό. Από τη μία είναι καταπληκτικό το ότι έχουμε τόσους ε, ικανούς ανθρώπους από τον τομέα της αλίας και ότι έχουν καταβληθεί τόσες προσπάθειες. Εάν είναι να συνεχίσει αυτή η κατάσταση και όχι να ε, επανέλθουμε στις δραστηριότητες του λόμπι, ε, ε, θα πρέπει να αλλάξει η δουλειά των ΡΑΚ. Δεν έχω εντολή από το ΡΑΚ της Βαλτικής να αναφέρω συγκεκριμένες θέσεις, επειδή την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση και θα έχω και άλλες τηλεφωνικές συζητήσεις Τέλη Δεκεμβρίου, λοιπόν, ίσως πριν τα Χριστούγεννα, θα μπορέσουμε να υποβάλουμε ε, σχετικό έγγραφο στην Κομισιόν. Αυτό σημαίνει ότι θα, θα μπορούμε να πούμε σαφώς πώς βλέπουμε ε, το μεταρρυθμισμένο ΡΑΚ και πώς βλέπουμε τα ζητήματα που, θα, ε, που αναφέρονται στην Πράσινη Βίβλο. Να πω όσον αφορά την Πράσινη Βίβλο ότι για πρώτη φορά βλέπω να υπάρχει τέτοια τιμιότητα από την κοινότητα. Η κοινότητα λέει ότι το σύστημα που έχουμε σήμερα δεν λειτουργεί. Θα πρέπει λοιπόν να μεταρρυθμίσουμε όλο το σύστημα. Και θα πρέπει επίσης να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να λαμβάνει υπόψη το νέο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ρόλο των ΡΑΚ και το ρόλο της Κομισιόν. Και αυτό δεν είναι απλό. Πιστεύω όμως ότι μπορεί να γίνει. το πρώτο θέμα που συζητήσαμε στο δικό μας ΡΑΚ και μιλάω μόνο για τη Βαλτική. Ξέρω πολύ καλά ότι κάποια ερωτήματα απατώνται διαφορετικά στα διάφορα ΡΑΚ. Θα μπορούσε να πει κανείς σχεδόν ότι η κοινότητα που δεν είχε κοινή αλληλευτική πολιτική. Οι προϋποθέσεις, οι συνθήκες είναι τόσο διαφορετικές ε, στις διάφορες περιοχές. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνούμε απόλυτα ότι παρότι υπάρχουν κάποια κίνητρα να αλλάξουμε την σχετική σταθερότητα που υπάρχει, ε, υπάρχουν πολύ ε, δύσκολα ζητήματα. Θα πρέπει να διατηρήσουμε το κομμάτι που, ε, για το οποίο αγωνιστήκαν με, επί 25 χρόνια στη Βαλτική. Ε, τα, κάθε κράτος δηλαδή να έχει αρμοδιότητες. Ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ελέγγυν και ε, αυτό ήταν το θέμα της πρώτης μάχης για τα ΤΑΚ. μπορούν ε, να γίνονται ε, ανταλλαγές ε, των ποσοστώσεων είτε μεταξύ κρατών είτε μεταξύ επιχειρήσεων. Συμφωνώ με όσους είπαν ότι θα πρέπει στη Βαλτική που έχει πολύ καλές προϋποθέσεις διότι συμμετέχουν λίγα κράτη-μέλη σχετικά θα πρέπει λοιπόν στη Βαλτική να υπάρχει μια σαφής κατεύθυνση από το ΡΑΚ, ε, να μην ε, συνεχιστεί η ε, διαρθρωτική πολιτική. Επίσης καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουν να συζητήσουμε μέτρα της αγοράς θα πρέπει να είναι δυνατόν όπως έχουν κάνει πολλά, πολλές χώρες να ε, σχεδιαστεί ένα σύστημα ποσοστώσεων το οποίο λαμβάνει υπόψη και τη βιολογία και την ε, αλία μικρής ε, κλίμακας. Δεν μπορούμε όμως να συζητάμε για ε, τις δομές, για την υπερβολική ικανότητα και να συζητάμε για χρήματα τη στιγμή που δεν λειτουργεί το σύστημα. Πιστεύουμε ότι η Βαλτική θα αποτελέσει κέντρο για κάποιου ε, είδους ε, ITQ, ενδεχομένως ε, στα πλαίσια του νέου συστήματος. Η, η, Πολωνία το συζητάει αυτό, η Δανία το έχει εφαρμόσει αυτό πλήρως, η Σουηδία το συζητάει. Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό. Διότι θα πρέπει να μειώσουμε την ικανότητα στην αλληλεία και θα πρέπει να καταλήξουμε σε αλληλεία νόμιμη και ε, που να ε, παρέχει αυτάρκεια στις χώρες. Ε, αλλά δεν είναι θέμα κιλοβάτ. Θέλουμε το Κοινοβούλιο να παρακολουθήσει ε, στενά το θέμα της μεταρρύθμισης των ΡΑΚ. Το θέμα είναι δεν να δημιουργήσουμε έναν μεγάλο γραφειοκρατικό μηχανισμό στα ΡΑΚ, αλλά κάποια ενίσχυση χρειάζονται. Για το ΡΑΚ της Βαλτικής είναι πολύ σαφές. ότι θα πρέπει να έχουμε ε, βοήθεια στο θέμα της ε, αξιολόγησης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αυτό. Δεν έχει να κάνει αυτό με τους βιολόγους της ICES, δεν έχει να κάνει με την ε, Κομισιόν. Κάποιος θα πρέπει να κάνει τη δουλειά αυτή, διότι Πολλοί κάνουν σαν να καταλαβαίνουν την αξιολόγηση αυτή, αλλά δεν την καταλαβαίνουν καθόλου ή, δεν καταλα... ή καταλαβαίνουν πολύ λίγα. Γιατί λοιπόν είναι αυτό τόσο σημαντικό στο μέλλον, διότι διότι η επαγγελματική αλία έχει συμβάλει πολύ λίγο στις παρούσες σχέσεις. Όλη η εμπειρογνωμοσύνη που υπάρχει θα πρέπει να σημαίνει ότι θα, θα μπορεί να υπάρχει πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Δεν θα πω σε λεπτομέρειε σχετικά με το ποιο θα πρέπει να είναι ο ενδιάμεσο φορέα ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στο ΡΑΚΑ. Αυτό που θα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Είναι πολύ σαφέ όμω ότι θα πρέπει να τονίσουμε ότι κάποια κράτη-μέλη ήταν ιδιαίτερα δραστήρια στα πλαίσια του δικού μα ΡΑΚ και άλλα όχι και επανειλημμένα έχω αναρωτηθεί πώς μπορεί να βελτιωθεί αυτό και πώς, ε, ε, ε, τι μορφή θα μπορούν να έχουν οι συνεισφορές των κρατών μέλων στα μέλλον. να σας ευχαριστήσω για την δυνατότητα να μιλήσω εδώ σήμερα και έκλεισε το μικρόφωνο του ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιωχάνσεν για 8 λεπτά στη συνέχεια. Έχει το λόγο ο κύριος ο οποίος ε, εκπροσωπεί το Περιφερειακό Συνόλιο Συμβουλίου των Όρκνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λέγομαι Λόρινο Κινέιντε. Και σε αντίθεση με τους συνδεύσεις είμαι πρόεδρος της, ε, Τουράκα ε, των Βορειοδυτικών Υδάτων. Εκπροσωπώ τον πρόεδρο. Κάνει κάτι που συχνά το ξεχνάμε. Ψαρεύει αυτή τη στιγμή και ζήτησε να σα μεταφέρω τη συγγνώμη του, διότι τη, να σα δει συγγνώμη γιατί δεν θα είναι παρόν. Καταρχήν, η παρουσίασή μου είναι προσωρινή, διότι το ράκ της περιοχής μου δεν ολοκλήρωσε τις, ε, τα συμπεράσματά του, αν και έχουμε μια εξαντλητική λεπτομερή διαδικασία προσπαθώντας να διατυπώσαμε τις απόψεις του ΡΑΚ σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της ΚΑΛΠ. Επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, το απαιτεί αυτό. Το ΡΑΚ των βορειοδυτικών υδάτων γεωγραφικά καλύπτει από τα δυτικά της Σκωτίας τα βόρειο-δυτικά της Σκωτίας μέχρι τη μάχη γύρω από την Ιρλανδία, την Αγγλία, αγγίζει τις ακτές της Γαλλίας. Είναι ένας μικρόκοσμος πολυπλοκότητας και διαφορές απόψεων. Λόγω αυτής της πολυμορφίας των μελών είναι μεγάλη πρόκληση στην απάντησή μας. Δεν θα απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα της Κομισιόν που ετέθησαν στην Πράσινη Βίβλο. Θα περιοριστούμε μόνο στα θέματα που τώρα αισθάνεται κάπως πιο άνετο στο να μπορεί να δώσει συμβουλή. Επειδή ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι πανευρωπαϊκοί οργανισμοί και εθνικά βήματα όπου θα σημειώνεται είσοδος στοιχείων στο σύστημα. Μόλις ο συναδέλφος των άλλων ΡΑΚ και εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει μεταρρύθμιση. Με βάση ορισμένες αρχές όπως ο συσχετισμός βιολογικών, οικολογικών συμφερόντων με οικονομικά. Μια από τις πιο μεγάλες δυσκολίες για την Αγία είναι η έλλειψη βεβαιότητας. Οι επιμέρους αποφάσεις είναι δύσκολες λόγω αυτού. και έχω μια γενικευμένη δυσφορία και απειλή για όλο τον κλάδο. Στο ΡΑΚ υπάρχουν διστάμενες απόψεις, παραδείγματος χάρη, για το αν πρέπει να κρατήσουμε τη χρήση των τάξ και των ποσοστώσεων ή να περάσουμε σε ένα άλλο σύστημα, όπου να γίνεται έλεγχος της προσπάθειας. Αυτό έχει σχέση φυσικά με την σχετική σταθερότητα. Και αυτό θα είναι, στο, θα το δείτε στο κείμενο που θα σας δώσουμε. Περιφερειοποίηση. Το ΡΑΚ είναι περιφερειακό όργανο. Άρα προορίζεται κατά κάποιο τρόπο υπέρ μιας περιφερειοποίησης πτυχών της ΚΑΛΠ όπως οι αποφάσεις να παίρνονται πιο κοντά στο σημείο επίπτωσης της απόφασης. Βέβαια υπάρχουν και όροι της συνθήκης που δίνουν στις κυβερνήσεις, την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο εξουσίες κεντρικές. Πώς λειτουργεί η περιφερειακή διάσταση. Η περισσότερο οι περισσότερε αφορούν τους φορεί βιομηχανικού και μη, επιστήμονες και κυβερνήσεις. Από πολύ νωρί, έτσι ώστε η κατάσταση να είναι σαφής ως προς το πώ θα ληφθούν οι αποφάσεις. Υπερβάλλουν δυναμικό στο στόλο. Δεν πρέπει να το υπεραπλουστεύουμε το θέμα αυτό. Πρέπει να ορίζουμε σωστά και να ελέγχουμε το μέγεθος του στόλου και το υπερβάλλον στοιχείο έτσι ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται δυνατόν κατά αλλιευτική μονάδα ή κατά χώρα. Επιστημονικά δεδομένα που στηρίζουν τις συζητήσεις μας όσον αφορά τη διαχείριση των αλλιευμάτων στα περισσότερα θέματα υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη αβεβαιότητα. Η νέα ΚΑΛΠ θα πρέπει να διαγράψει μια πορεία όπου η άρση αυτής της αβεβαιότητας να ορίζεται διαχρονικά. Γιατί και περιβαλλοντικά και αλλιευτικά δεν έχει νόημα να παραμένει αυτή η αβεβαιότητα γύρω από μεγάλες αποφάσεις. Θέλουμε έλεγχο, αναθεώρηση στην αρχή μιας τέτοιας διαδικασίας έτσι να ορίζεται αν χρειάζεται να αλλάξει η μεθοδολογία διαφοροποιημένη διαχείριση. Αυτό γενικά το επικροτούμε, μόνο που θα πρέπει να γίνει σαφής εξέταση του πολύπλοκου χαρακτήρα του θέματος αυτού. Η αλία μπορεί να είναι απλή, αλλά η διαχείριση της αλίας είναι σύνθετη. Δεν υπάρχει μία λύση για όλα και για όλους. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, το θέμα της αγοράς και της χέρις μεταξύ της διαχείρισης των αλλιευμάτων, της εμπορικής πολιτικής και της πολιτικής περιβάλλοντος πρέπει να το δούμε μες στα πλαίσια της μεταρρυθμισμένης αλλιευτικής πολιτικής γιατί δεν μπορούμε να έχουμε αρχές που να ισχύουν για την κοινοτική αλληλεία και το κοινοτικό περιβάλλον και να μην εφαρμόζονται στους ανταγωνιστές μας. Θα σας στείλουμε γραπτά τα απορίσματά μας και σε εσά και στην Κομισιόν πριν τα Χριστούγεννα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να το στείλετε εγγράφος. Ευχαριστώ κύριε Οκινέιντε. Στη συνέχεια δίνω το λόγο στον ε, κύριο Καμπράλ. 8 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την προσωπική σας ε, πρωτοβουλία για τη διοργάνωση αυτής της ακρόασης και την διαθεσιμότητά σας να ακούσετε τις απόψεις όλων σε σχέση με τη νέα αυτή αλληλευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πέντε κύρια κεφάλαια σε ό,τι αφορά την κοινή αλληλευτική πολιτική. Καταρχήν έχουμε τους στόχους για την εξωτερική διάσταση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής την περιφερειακή διαχείριση με οργανισμούς, τις αλληλευτικές συμφωνίες, το εμπόριο, τις αγορές και την μεταποίηση. Επίσης, τρίτον, διακυβέρνηση και ευθύνη, τέταρτον, τη διαρθρωτική πολιτική και πέμπτον, τα επιστημονικά στοιχεία. Η τωρινή αλληλευτική πολιτική δεν ήταν σε θέση να επιλύσει τα κύρια προβλήματα του αλληλευτικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η υπερβολική εκμετάλλευση, η υπερβολική αλληλευτική ικανότητα, οι μεγάλες ενισχύσεις και τη μείωση των αλληλευτικών πόρων. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το σωστό στόλο για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Πρέπει να υπάρξει μια ανάλυση η οποία θα λάβει υπόψη το ρόλο όλων των φορέων και των παίκτων. Το LDRAC δεν συμφωνεί πλήρως με την ανάλυση η οποία έχει παρουσιαστεί από την Κομισιόν στην Πράσινη Βίβλο ούτε με μερικές από τις κατευθύνσεις και τους προσανατολισμούς που προτείνονται εκεί. Ο, ο συνολικός στόχος μας θα πρέπει να είναι να προωθήσουμε την υπεύθυνη και αηφόρο αλληλεία στον τομέα του περιβάλλοντος, τον κοινωνικό και τον κοινωνικό τομέα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να εξασφαλίσουμε μια ανταγωνιστική και κερδοφόρα αλληλεία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το στόχο της τροφοδότησης και της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αυτός ο στόχος πρέπει να τύχει συντονισμού με άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να είναι και συνεκτικός με τον στόχο της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν τρεις κύριοι τομείς εξωτερικής διάστασης της κοινή πολιτικής, όπως σας είπα. Οι περιφερειακοί οργανισμοί για τη διαχείριση των αλληλεγμάτων. είναι ένα πλαίσιο με στο οποίο υπάρχει διαχείριση των διεθνών υδάτων, οι εταιρικέ συμφωνίε αλίας και τρίτον τα θέματα εμπορίου, αγορών και μεταποίηση. Σε ό,τι αφορά το πρώτο φορέα, του περιφερειακού φορεί, <clears throat> η έλλειψη ενδιαφέροντος για την αλία σημαίνει και έλλειψη πολιτικής επιρροής. Η κοινή αλληλευτική πολιτική πρέπει να προωθήσει την ε, αηφόρο διαχείριση των αλληλευτικών δραστηριοτήτων μέσω της συμμόρφωσης και της καλής διαχείρισης και της ευκυβερνησίας του τομέα. Πρέπει επίσης να εξεύρει μια ισορροπία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στους φόρους και ένα σύστημα το οποίο θα είναι διάφανο και δεν θα έχει διακρίσεις. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στη συμμόρφωση γιατί αυτή και είναι και η βάση για τις απαραίτητες επιστημονικές μελέτες που θα οδηγήσουν τα κατάλληλα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Η εναρμόνιση των περιφερειακών φορέων διαχείρισης είναι απαραίτητη επίσης σε ό,τι αφορά τα οριζόντια θέματα. Σε ό,τι αφορά τις εταιρικέ σχέσεις και συμφωνίες για την αλία, είναι η δεύτερη γενιά συμφωνιών που έχουμε με τρίτες χώρες, η κοινή αλληλευτική πολιτική θα πρέπει να παροτρύνει <clears throat> την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω χρηματοδότησης για να βελτιωθούν οι τεχνικές προδιαγραφές της εφαρμογής των συμφώνιων αυτών, να, να βελτιωθεί το επίπεδο της συμμετοχής των εμπλεκομένων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, να εξασφαλιστεί η εδρεωμένη επιστημονική γνωμοδότηση, να υπάρξει ευκυβερνησία και διαφάνεια και να προωθήσουμε ένα κλίμα συμμόρφωσης. Η περιφερειακή προσέγγιση για την ευκυβερνησία όμως μόνο σε ορισμένες περιοχές μπορεί να εφαρμοστεί. Θα πρέπει να έχουμε μια διάκριση μεταξύ του κόστους πρόσβασης για τον στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μακρών αποστάσεων που να καλύπτονται από τους εφοπλιστές και την χρηματική συμμετοχή της κοινή αλληλευτικής πολιτικής σε ό,τι αφορά την εξάλληψη της ένδυας και την ανάπτυξη. Καλές συμφωνίες οι οποίες δεν έχουν πραγματικές δυνατότητες αλίας θα μπορούσαν να θεωρηθούν σαν μέσο πρόθεση συνεργασία των επενδύσεων και των κοινοπαξίων με τρίτε χώρε. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και τα περιφερειακά συμβούλια οργάνωση και οι αλληλευτικέ συμφωνίε θα πρέπει να έχουν περισσότερου ανθρώπινου πόρου και να δοθούν και αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη για καλύτερη διαχείριση του διοικητικού άχθους εφαρμογής τους. Οι αγορές και η μεταποίηση. Η ανάλυση στην Πράσινη Βίβλο είναι απλοϊκή και πολλές φορές αντιφατική. Δεν λάμβανε υπόψη τον κύριο ρόλο που πέσουν αυτά τα στοιχεία για την επίτευξη των συνολικών στόχων της κοινής αλληλευτικής πολιτικής. Η συμμετοχή της μεταποιητικής βιομηχανίας για τα αλλιεύματα δεν λαμβάνεται υπόψη επίσης επαρκώς στην ανάλυση του μέλλοντος κοινής ε, αλληλευτικής πολιτικής. Οι συμφωνίες για πρόσβαση στην αγορά είναι ένα βασικό στοιχείο των συμφωνιών στον βόρειο χώρο για τα θέματα αυτά και μιλώ ιδιαίτερα για την Ορβηγία που είναι ένας ιδιαίτερος εταίρος μας. Έρχομαι στην εμπορική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει την αηφόρο και υπεύθυνη πολιτική αλίας και μια αποτελεσματική εμπορική πολιτική που θα εξασφαλίσει η ισορροπημένη προμήθεια της αγοράς της Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να εξασφαλίσει ότι έχουμε ένα ισόπεδο γήπεδο σε ό,τι αφορά την αλία και τα αλληλευτικά προϊόντα είτε είναι ευρωπαϊκά είτε εισαγόμενα σε σχέση με την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων σε επίπεδο παραγωγής, μεταποίησης και τελικού προϊόντος. Οι συνθήκες πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο για την αηφόρο, θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο για την αηφόρο αλία. Είναι απαραίτητο να υπάρξει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα σε όλα τα στάδια της αλίας μέσω των διεθνών φορέων και της οργάνωσης αλίας με την ανάπτυξη των καταλήλων ελέγχων ώστε να τηρούνται οι κανόνες της αγοράς. Να υπάρξει και μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα και την ανάπτυξη στον τομέα της αλίας. Να υπάρξει ένας μηχανισμός διαφάνειας για να φαίνονται και οι διαφορές μεταξύ τιμής κόστους και τιμής τελικής για τον καταναλωτή. Βελτίωση της διαφάνειας για να υπάρχουν νέοι και για, για τους νέους κανονισμούς να λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την άποψη όλων των εμπλεκομένων στην αγορά. Έμφαση επίσης να δοθεί όχι μόνο στις, αγορές, στις τιμές, αλλά και στο κόστος παραγωγής και μεταποίησης. Είναι απαραίτητο επίσης να υπάρξει διακυβέρνηση και ευθύνη. Θα πρέπει να έχουμε μια εκ των κάτω λήψη αποφάσεων και όχι όπως είναι τώρα εκ των άνω προς τα κάτω. Δηλαδή να φύγουμε από την κεντροποιημένη και μικροδιαχειριστική προσέγγιση. Θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι στα τοπικά ΡΑΚ να είναι σε διαπραγματεύσεις των κρατών μελών με τρίτες χώρες. Αυτό θα βελτιώσει τις διαπραγματεύσεις αυτές και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξέρει τους κατάλληλους μηχανισμούς για να λάβει υπόψη την άποψη όλων των εμπλεκομένων κατά τη διάρκεια της ε, διαπραγματεύσης διαρθρωτική πολιτική. Οι στόχοι θα πρέπει να τίθενται σε συνάρτηση με την κοινή, αγροτική πολιτική, κοινή αλληλευτική πολιτική. Οι μηχανισμοί θα πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να υπάρχει ένα σύστημα για τη διαχείριση των πόρων του εξωτερικού στόλου που να συμβαδίζει με τα σχέδια τα οποία έχουν ε, γίνει δεκτά για τον τόνο και την ε, αηφόρο ανάπτυξή του. Για την επιστημονική επίση εμπειρογνωμοσύνη είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι ανεξάρτητε μελέτε και θα, υπάρξει, θα πρέπει να υπάρξει εστίαση σε ειδικέ μελέτε για την υπερβολική αλληλευτική ικανότητα. Οι δράσει πρέπει να λαμβάνονται από τη βάση ε, εδρεωμένων επιστημονικών απόψεων και μόνιμη επαφή με του εμπλεκομένου στον τομέα αυτό για να βελτιωθεί η ποιότητα αυτών των γνωμοδοτήσεων. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καβράλ ακολουθεί για 8 λεπτά ο πρόεδρος των πελαγικών ΡΑΚ, ο κύριος Μαξουίν. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για τη δυνατότητα αυτή να, συμμετέ... να συμμετάσχω στη συζήτηση σήμερα. Εδώ και κάποιο καιρό αναγνωρίζεται γενικά ότι το θεσμικό πλαίσιο γύρω από την κοινή αλλιευτική πολιτική έχει κάποιες ελλείψεις. Και η τελευταία αναθεώρηση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής ε, έδειξε ότι μια από τις βασικές ελλείψεις ήταν η έλλειψη της ε, συμμετοχής των διαφόρων ενδιαφερομένων στη διαδικασία. Αυτό οδήγησε στη δημιουργία των ε, Περιφερειακών Συμβουλίων, των ΡΑΚ, που εκπροσωπούνται εδώ σήμερα. Στο πελαγικό ΡΑΚ πάντα θεωρούσαμε την ε, δημιουργία μας ε, ως ε, εξελικτική διαδικασία. Η πιο βασική η πιο βασική λειτουργία στην μπορούμε να συμμετάσχουμε είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα πελαγικά ψάρια και εποφελούμαστε από τη συνεργασία των μη κυβερνητικών οργανώσεων, διότι επειδή αναφερόμαστε όλο και περισσότερο στην, ε, ε, ε, στην διαπίστευση και στην ανιχνευσιμότητα, είναι σημαντικό οι μη κυβερνητικέ οργανώσει να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία. Ε, κυρία Πρόεδρε, εγώ αυτό που θέλω να σα πείσω όμω είναι ότι η, πελαϊκή αλληλεία είναι διαφορετική. Θα ήταν ωραίο να δημιουργήσουμε μια πολιτική η οποία να εφαρμόζεται σε όλε τι περιπτώσει. Εάν δείτε όμω τον κατάλογο των ράκ που εκπροσωπούνται εδώ σήμερα, με εξαίρεση το πελαγικό ρακ, όλα τα άλλα είναι περιφερειακά. Και αυτό φαίνεται από τον τίτλο τους. Η δυσκολία του δικού μας τομέα είναι ότι τα πελαγικά είδη δεν γνωρίζουν σύνορα. Όπως ε, η Πεσκαδρίτσα για παράδειγμα ε, την βρίσκουμε από τον Νότιο Ατλαντικό μέχρι την, ε, μέχρι την ακτική Το πρόβλημα που δημιουργείται λοιπόν κυρία Πρόεδρε είναι ότι για μέρος της μεταναστευτικής τους πορείας τα ψάρια περνάνε από ύδατα χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιφερειακά συμβούλια ασχολούνται με τα προβλήματα της περιφέρειάς τους, ε, αλλά ε, στη δική μας περίπτωση κάποιες περιφέρειες ε, δεν ανήκουν σε εμάς και γι' αυτό χρειαζόμαστε κάπως διαφορετική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις και στη δημιουργία πολιτικής. Είναι πολύ λυπηρό ότι για κάποια είδη, κάποιες χώρες όπως η Ισλανδία, μπορούν να ανακοινώσουν ότι σκοπεύουν να ε, αλλιεύσουν 130.000 τόνους ε, σκουπρί παραπάνω του χρόνου. Ή ότι οι Νορβηγοί φέτος ε, θα αλλιεύσουν 100.000 περισσότερους τόνους αφρίδια. Η βιώσιμη αλλιευτική πολιτική υπονομεύεται από την ικανότητα εξωτερικών ε, εταίρων να λάβουν ε, μονοπλευρές αποφάσεις ε, σχετικά με την διαχείριση των αλλιευμάτων. Και για τον λόγο αυτό βρίσκομαι στην κάπως περίεργη θέση, να πω, ως πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου να ζητώ από το Κοινοβούλιο να είναι προσεκτικό όσον αφορά την περιφερειοποίηση της αλίας, διότι μέχρι να συναντήσουμε το πρόβλημα της αντιμετώπισης των τρίτων χωρών που συμμετέχουν στην αλία αυτή, στον πελαγικό τομέα θέλαμε ε, συγκεντρωμένη αποκεντροποίηση, διότι χρειάζεται ένας ισχυρός εταίρος που να μπορεί να διαπραγματευτεί με τις χώρες αυτές. Είναι σημαντικό λοιπόν να έχουμε αυτή την προσέγγιση. Κυρία Πρόεδρε, αναφερθήκατε στην, στο πρόβλημα των απορρίψεων. Να είμαι ειλικρινή. η διαχείριση των, της πελακής είναι μάλλον ε, ευκολότερη από ό,τι για τα άλλα είδη, διότι αν ε, κάποιος αλλιεύει ένα είδος, συνήθως δεν έχει πρόβλημα απόρριψης. Ε, μπορεί να έχει πρόβλημα διαβάθμισης, αλλά αυτό είναι διαφορετικό θέμα. Εμείς στο δικό μας ΡΑΚ πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα με την παρακολούθηση των εκφορτώσεων, διότι εάν απορρίπτει κανείς όλα τα μικρά ψάρια και εκφορτώνει τα μεγάλα, αυτό ε, θα φανεί πολύ γρήγορα στην αγορά. Αλλά στο δικό μας πλαίσιο, κυρία Πρόεδρε, αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος της αλληλευτικής προσπάθειας δεν είναι κατάλληλο εργαλείο για τη διαχείριση των πελαγικών ειδών τα πελαγικά, η πελαγική αλία ε, επικεντρώνεται σε αλλιεύματα τη στιγμή που έχουν την υψηλότερη ποιότητα και μπορούν να πετύχουν τις υψηλότερες τιμές στην αγορά. Ε, κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν, διαφορέ διαφορές ανάμεσα στα είδη και έχω κατανόηση για το έργο σας που προσπαθείτε να συνδυάσετε τις διάφορες πτυχές ε, όχι μόνο όσον αφορά τα μεμονωμένα είδη απέναντι στα μεικτά αλλά και την βιομηχανική αλία με τη βιοτεχνική αλία. Είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί η ισορροπία αυτή. Θα πρέπει όμως να την πετύχουμε. Μπορεί η λύση στον Βόρειο Ατλαντικό να είναι να πείσουμε την Νορβηγία και τις Φερόες νήσους να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι αυτό ε, θα μας δώσει τη βάση για περιφερειακή διαχείριση. Αλλά ε, όσο όλα πρόκειται το κοινοβούλιο σας μάλλον θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτό σύντομα. Πάντως είναι ενδιαφέρον που βλέπουμε ότι προχωράει η προσχώρηση της ε, Ισλανδίας και θα παρακολουθήσουμε ενδιαφέρον τις διαπραγματεύσεις ε, με την Ισλανδία στον τομέα της αλληλείας. Κλείνοντας, ε, φοβάμαι ότι το μήνυμα που προσπαθώ να σας μεταφέρω είναι ότι η πελαγική αλληλεία αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει μία λύση για, όλες, για όλα τα αλληλεύματα. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι στα πλαίσια της επίτευξης ε, μακροπρόθεσμων ε, σχεδίων αλληλείας και βιώσιμης αλληλείας, ε, ο μόνιμος διάλογος μεταξύ των ενδιαφερομένων έχει να παίξει σημαντικό ρόλο και μάλιστα διάλογος όχι μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με τους εταίρους μας από τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό κυρία Πρόεδρε, στις ε, συνεδριάσεις μας αναφέρεται συχνά το ότι τα, πόσο ενοχλητικό είναι το ότι τα πελαϊκά είδη ε, χρησιμοποιούνται για να επιτευχθούν συμφωνίες με τρίτες χώρες. Θα θέλαμε να μπορούμε να αλλιεύουμε τα πελαγικά είδη εντός των υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαξουίν. Για να κλείσουμε με τα περιφερειακά συμβούλια και το ΡΑΚ της Μεσογείου δεν έχει απαντήσει στην πρόσκλησή μας, γι' αυτό δεν είναι παρόν στην ακρόαση αυτή. Για να κλείσουμε λοιπόν ο κύριος Μπαριόλα, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του ΡΑΚ των ε, νοτιοδυτικών υδάτων. Συγγνώμη, θα σας δώσω μετά το λόγο. Ο κύριος Μπαριόλα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να μπορέσω να εκφράσω την άποψη του ΡΑΚ των Νοτίων Ιδάτων, που είναι η περιφερειακή οργάνωση όπου έχει την πιο μεγάλη σημασία ο βιοτεχνικός ή αλλιευτικός στόλος. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για να το έχετε υπόψη γιατί δεν καλύπτουμε μονάχα μια ευρεία γεωγραφική περιοχή, αλλά έχουμε και ιδιαίτερες πτυχές κοινωνικές και πολιτιστικές στο δικό μας Περιφερειακό Συμβούλιο. Ξεκινώ από ένα βασικό από το βασικό αυτό στοιχείο ότι θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την σκέψη που αποδίδει η Πράσινη Βίβλος στην κοινή αγροτική, κοινή αλληλευτική συγγνώμη, πολιτική. Και πρέπει να πούμε ότι μέχρι στιγμή η διαχείριση και η διακυβέρνηση αυτού του τομέα ήταν μια απόλυτη αποτυχία γιατί ήταν απόλυτα άκαμπτη η διαχείριση αυτή. Και γι' αυτό τονίζουμε την ανάγκη να υπάρξει μια περιφερικοποιημένη διαχείριση. Στην περίπτωση του δικού μας ΡΑΚ έχουμε τρεις περιοχές οι οποίες μπορούν να έχουν κοινή αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά τους ε, ε στόλους τους. Έχουμε τον ε, στόλο του κόλπου της, ε, το Βισκαϊκό, έχουμε τον στόλο των Ιβυρικών θαλασσών και επίσης έχουμε τον στόλο της περιοχής το, της Μαδέρας και των Καναρίων. Σε ό,τι αφορά στους στόχους, εγώ θέλω να υποστηρίξω την, υπο, την μείωση των απορρίψεων. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι μέσα σε αυτή την τάση υπάρχει και ένα είδος ε, σιωπής από την πλευρά της Κομισιόν που δείχνει ότι η Κομισιόν δεν θέλησε να αντιμετωπίσει σε όλη την έκτασή της το πρόβλημα αυτό των απορρίψεων γιατί υπάρχουν και απορρίψεις ορίμων ηχθείων που έχουν εμπορική αξία λόγω εξάντλησης των ποσοστώσεων. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακόμα και αν πρέπει να λάβουμε υπόψη την αρχή της σχετικής σταθερότητος σε ό,τι αφορά την ε, αγορά. Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να έχουμε μία αηφορία χωρίς να εξασφαλίσουμε πραγματικά ανεκτά εισοδήματα στους αλείς. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τους Ευρωπαίους αλείς εγκαταλελειμμένους σε μία αγορά η οποία είναι μια ζούγκλα όπου υπάρχει τεράστια επιθετικότητα, όπως υπάρχουν προϊόντα τα οποία προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν υπάρχει καμία απέτηση καμιάς προδιαγραφής ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική ευθύνη, την, ε, ε, τον έλεγχο της ποιότητάς τους κτλ. Είμαστε τελείως επομένως στο έλεος αυτών των ξένων αλλιέων. Θα πρέπει να έχουμε μια, ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέψει να επιβιώσει η ευρωπαϊκή αλληλεία σε ένα επίπεδο αξιοπρέπεια. Σε ό,τι αφορά την χωροταξία και την αντιμετώπιση των διαφόρων μορφών αλίας, εμείς επειδή έχουμε ένα ισχυρό χαρακτήρα σε ό,τι αφορά την βιοτεχνική αλία, δεν μπορούμε να έχουμε ιδιαίτερη γνώμη σε ορισμένα θέματα, όπω παραδείγματο χάρη η πρόσβαση πέραν των 12 μιλίων. Γιατί ο Βιοτεχνικό στόλο θα πρέπει να έχει μια τελείω διαφορετική αντιμετώπιση. Δεν θεωρούμε όμως ότι πρέπει να είναι αποκλειστικό ο έλεγχος η πρόσβαση στα 12 μίλια από τον βιοτεχνικό στόλο. Και επίσης εμείς δεν υποστηρίζουμε το να υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι θα εκφεύγουν από τον έλεγχο των κρατών μελών θέλουμε να τονίσουμε ότι υπάρχει μια σημαντική διαφορά σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση από το δικό μας Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε λοιπόν ένα στόχο ο οποίος δεν θέλει να τροποποιηθεί η αρχή της σχετικής ε, σταθερότητας, ο δε στόλος ανοιχτής θάλασσας θέλει να εξασφαλίσει μια ευκαμπτοποίηση της, ε, της ε, σχετικής σταθερότητας μέσω συμφωνιών κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά τις επιστημονικές γνώσεις, δεν ξέρω ότι αν εδώ θα έπρεπε να μιλήσω για μομφή, αλλά πρέπει να πω ότι μια πρωτοβουλία η οποία έχει παρουσιαστεί από το Συμβούλιο του Νότου, το σχέδιο ΧΕΠΕΤΟ, δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη στις πρόσφατες συνεδριάσεις. Ξέρουμε γιατί, γιατί εμείς θεωρήσαμε ότι δεν ελήφθη υπόψη σοβαρά ένα σχέδιο των διαστάσεων που έχει το ΧΕΠΕΤΟ που εμείς θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να είναι ένα υπόδειγμα για το μέλλον, ένα υπόδειγμα για μακροχρόνια διαχείριση. Είναι οδυνηρό το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος της Κομισιόν στην ε, κυβέρνηση της χώρας την οποία ενδιαφέρει ιδιαίτερα το πρόγραμμα αυτό δεν ήξερε καν τι είναι τα ΡΑΚ, τα Περιφερειακά Συμβούλια. Αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο μας φαίνει σε απόγνωση. Πώς μπορούμε λοιπόν να έχουμε μια στοιχειώδη απήχηση μέσα στην γραφειοκρατία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από τέτοιες συνθήκες. Τώρα, ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Η αλληλεία βρίσκεται εγκαταλελειμμένη στη δίχη της πολύ συχνά και κανείς δεν σκέφτεται τα θέματα της χρήσης του, των θαλασσών και του θαλασσίου χώρου, παρά το γεγονός ότι είναι μια πολύ παλιά δραστηριότητα η αλία και το γεγονό ότι οι αλίε έχουν μια πολύ καλύτερη γνώση των θαλασσών από του άλλου χρήστε βρίσκονται σε εγκατάλειψη γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν επιρροή. Στην, ε, στον καθορισμό των δραστηριοτήτων στη θάλασσα θέλουμε όλε αυτέ τι δραστηριότητε που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα να έχουν επιστημονική βάση και να αφήνουν επαρκή χώρο στην θαλάσσια, στην ε, θαλασσία Θέλουμε επίσης να υπάρξει μια ομογενής ε, συγκέντρωση δραστηριοτήτων για να μην υπάρχει μια μονομερής μονάχα διαχείριση των θαλασσών χωρίς να λαμβάνει υπόψη την αλία. Τέλος, θέλω να τονίσω σε σχέση με την βιοτεχνική αλία ότι είναι απαραίτητο να την υποστηρίξουμε, να συνεχίσουμε τις ενισχύσεις και να εξασφαλίσουμε ότι θα εξακολουθήσει να υπάρχει βιοτεχνική αλία στις θάλασσες του Νότου. Ευχαριστώ. Μονάχα να σας πω ότι εμείς αγωνιζόμαστε η θαλάσσια πολιτική και η αλληλεία να συνδυάζονται και η αλληλεία να παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή την θαλάσσια πολιτική. Αυτό είναι ακριβώ ένα κοινό αγώνα και εμεί αγωνιζόμαστε για το θέμα αυτό από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριο Γιάννη, που ζήτησε τον λόγο και μετά θα έχουμε τη συζήτηση. Κύριε Γιάννη. Ε, no. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέγομαι Γιάννη και είμαι αντιπρόεδρος του ΡΑΚ και με επιφόρτησε ο πρόεδρος να σας μεταφέρω τη φωνή του Μεσογειακού ΡΑΚ. Μετά θα πρέπει να, ε, να μιλήσω ως ε, ε, πρόεδρος της Λέγκα Πέσκα. Για να μην μιλήσω δύο φορές, θα μπορούσα να μιλήσω μία αν μου επιτρέπετε. Πρόεδρος. Όχι, όχι. Αυτό το οποίο θα σας πω ως πρόεδρος της Επιτροπής αυτής, ότι το ΡΑΚ της Μεσογείου δεν έδωσε απάντηση παρά το γεγονός ότι προσεκλήθη. Θα έχετε τη δυνατότητα να λάβετε το λόγο το απόγευμα. Αλλά εγώ δεν έδωσα κάποια, κάποιο σχόλιο για το ράκ της Μεσογείου. Απλώς ότι προσεκλήθη αλλά δεν απάντησε και εσείς ερχόσαστε με ένα άλλο καπέλο ούτως υπήν. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν όλους αυτούς οι οποίοι έχουν λάβει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε σεβαστεί τον χρόνο αγόρευσης γιατί έχουμε μονάχα μισή ώρα για τη συζήτηση που πρέπει να επακολουθήσει θέλω να ζητήσω από όλου αυτού οι οποίοι θα λάβουν το λόγο να μην κάνουν να μην εκφωνήσουν λόγους, αλλά να κάνουν ερωτήσεις, οι οποίες μπορούν να απαντήσουν οι προσκεκλημένοι μας. Και δίνω καταρχήν το λόγο στον κύριο Στίβενσον. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ενδείκνυται, όπως είπατε, να γίνεται αυτή η ακρόαση την 1η Δεκεμβρίου, γιατί η συνθήκη της Λισαβόνας μας δίνει εξουσίες απόφαση. Άρα είναι σωστή η ημερομηνία αυτή. Όμως, κάτι που ακούσαμε από πολλούς με σαφήνεια είναι ομοφωνία εκ μέρους όλων ότι μία λύση για όλους δεν είναι η σωστή μέθοδος. Αυτό δοκιμάστηκε εδώ και 29 χρόνια και απέτυχε. Μικροδιαχείριση εκ μέρους των Βρυξελών υπήρξε αποτυχία. Σημειώνω αυτά που είπε ο Ιαν Σουίνγκ. Δηλαδή, δεν πρέπει να βιαστούμε. Να έχουμε μια αποκεντρωμένη πολιτική με ένα σύστημα μία λύση για όλους και πάλι. Η συγκέντρωση απέτυχε αλλά και η αποκέντρωση θα αποτύχει αν πάμε να δώσουμε μία μέθοδο εκ των άνω λύσης. Bottom down. Θα πρέπει να αφήσουμε τα διαχειριστικά συστήματα στα κράτη-μέλη. Συμφωνώ με αυτή την άποψη. Γιατί είναι τόσο μεγάλες διαφορές υπάρχουν στην Αγγλία μέσα στην Ένωση και όπως είπε ο Ιαν Μαξίν και πάλι ιδιαίτερα στα πελάγια είδη ώστε θα πρέπει την καθημερινή διαχείριση αν θέλουμε και όλοι οι φορείς, οι επιστήμονες, οι αγγείες να παίρνουν όλοι μέρος, θα πρέπει να αφήσουμε τις κυβερνήσεις να αποφασίσουν ποιο είναι το καλύτερο για αυτές. Στι Βρυξέλλες θα έχουμε την κοινή ελληνική πολιτική. Θα είμαστε ο τελικός διαιτητής. Να δούμε ότι να φροντίζουμε να υπάρχει διατήρηση των αποθεμάτων και να εφαρμόζονται οι κανόνες σωστά αλλά ο περιορισμός της προσπάθειας αν θα είναι η καλύτερη απόφαση για, την, για τα μεικτά αλλιεύματα, ναι. Αλλά όχι όμως για τα ίδια ανοιχτή θαλάσσης, όπου θα πρέπει να συνεχίσουμε, όπως γίνεται μέχρι τώρα, με τα τάξη και τις ποσοστώσεις. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε την πολυμορφία, να αντιλάβουμε υπόψη μας. Επίσης, θα ήθελα και του είπε η συγγήτρια να τονίσουμε ιδιαίτερα τις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Ταυτόχρονα όμως να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε και νησιωτικές περιφερειακές μεγάλων αποστάσεων ως προς τις υπόλοιπες κοινότητες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή όπως ε, τα νησιά Σέτλαντ. Πρέπει και σε αυτό να δοθεί έμφαση. Ελπίζω να ληφθεί υπόψη αυτό από του εισηγητές μα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βαλέσα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα της περιφερικοποίησης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο τίθεται και από την Πράσινη Βίβλο για την Πολωνία και τη Βαλτική. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί έχουμε και μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό αυτή τη στιγμή. <clears throat> Υπάρχει ένα συμβουλευτικό συμβούλιο ΝΑΡΑΚ τη Βαλτικής και υπάρχουν και οικολογικέ οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια του και το Συμβούλιο αυτό έχει δώσει την άποψή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΜΕΝ, αλλά αυτή τη στιγμή ελείπουν τα στοιχεία που θα μα επιτρέπουν να γνωρίσουμε ποια είναι η σύνδεση μεταξύ του ΡΑΚ αυτού και των ε, αλευτικών φορέων των χωρών της Βαλτικής. Στη Στοκχόλμη πρόσφατα με πρωτοβουλία της ε, Σουηδικής Προεδρίας υπεγράφει μια συμφωνία για την αλληλεία στη Βαλτική. Το κείμενο αυτό περιλαμβάνει και μια πρόταση για να δημιουργηθεί ένα περιφερειακό όργανο, ένα είδος στρογγυλής τραπέζης για την αλληλεία στην ε, Βαλτική που θα περιέχει, θα περιλαμβάνει μάλλον και το ΡΑΚ και τις εθνικές διοικήσεις για την αλληλεία στις χώρες Βαλτικής και επιστήμονες επίσης. Βέβαια, αυτό οδήγησε σε επικρίσεις και των αλλιέων σε σχέση με το γεγονός ότι το όργανο αυτό δεν προβλέπει την περιφερικοποίηση. Ποια είναι η άποψη της Κομισιόν λοιπόν για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο, η κυρία Λέβιν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον που ακούσαμε ότι υπάρχει σχετικά μεγάλη ε, συνένεση. Το θέμα της περιφερειοποίησης επανέρχεται συνεχώς. Σημείωσα ότι αρκετοί ανέφεραν ότι από την Πράσινη Βίβλο λείπει η κοινωνική διάσταση και νομίζω ότι είναι φυσικό να τονίσουμε σήμερα το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε έναν ε, καλό τομέα αλίες. Η κοινωνική ασφάλεια ε, αποτελεί συνέπεια αυτού. Υπάρχουν όμως πολλοί ενδιαφερόμενοι στον τομέα αυτόν, όχι μόνο οι επαγγελματίε αλληλεί, αλλά και ε, οι καταναλωτές, ε, οι φίλοι του περιβάλλοντος κλπ. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Όσον αφορά την συνάντηση στην Κουρούνια, που ε, θα έχει ω θέμα την αλλιευτική πολιτική, και το κοινό, μη κυβερνητικέ οργανώσει θα συμμετάσχουν ή μόνο επαγγελματικέ οργανώσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήταν χρήσιμο που ακούσαμε από ανθρώπους που ξέρουν, που γνωρίζουν το ζήτημα τώρα που συζητάμε την ε, μεταρρύθμιση του, της κοινή αλλιευτικής ε, πολιτικής. Νομίζω ότι αναφέρθηκε επανειλημμένα το ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει μία λύση για όλους. Χαίρομαι που ο κύριος Στίβενσον ε, συμφωνεί με αυτά που είπα εγώ χθες στην Επιτροπή. Ότι δηλαδή άμα είναι να καθόμαστε εδώ πέρα όπως κάνουμε τακτικά και φαίνεται να συμφωνούμε ότι η αποκέντρωση είναι καλή ιδέα, δεν θα πρέπει να ξεκινήσουμε την προσέγγιση μας στο θέμα της μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτικής πολιτική με την αποκέντρωση στην κορυφή των προτεραιοτήτων μα ε, και όχι στο τέλος ε, αφού ασχοληθούμε με το ε, ποιες διαχειριστικές δομές μπορούν να συμφωνηθούν σε κεντρικό επίπεδο. Νομίζω λοιπόν ότι τα όσα ακούσαμε σήμερα συμφωνούν με αυτά που ακούω εγώ στην πατρίδα μου, ότι θα πρέπει να κινηθούμε προς ένα σύστημα όπου τα κράτη που έχουν αλλιευτικά δικαιώματα σε διάφορες περιοχές όπως η Βόρεια Θάλασσα ή για πελαγικά είδη θα πρέπει να είναι αυτές που λαμβάνουν τις αποφάσεις σχετικά με το πώς θα γίνεται η διαχείριση των αλλιευμάτων αυτών στο μέλλον. Ο κύριος Μαξουίν, πολύ σωστά, ανέφερε την ανάγκη να συμμετάσχουν η Ισλανδία, η Νορβηγία και οι Φερόες Νήσεις στις ε, διαπραγματεύσεις. Είναι αξιοζήλευτη η θέση των χωρών αυτών. Η Νορβηγία στις ετήσιες συζητήσεις ε, ε, επηρεάζει, έχει, έχει μεγαλύτερο βάρος στη συζήτηση για την κοινή αλληλευτική πολιτική από ό,τι έχει το δικό μου κράτο μέλο η, το, η περιοχή από, από που έρχομαι εγώ, η Σκωτία. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Γενικό Διευθυντή. Ε, πριν κάποιες εβδομάδες ε, έγινε μια συζήτηση με τον Επίτροπο Μπόρε και ρωτήθηκε τι θα μπορούσε, ε, με, τι μέσα θα μπορούσαμε να, να ε, προσελκύσουμε την ε, Ισλανδία. Και ο Επίτροπος Μπόζ ε, ανέφερε μια λύση που εφαρμόστηκε για, την, για το δικό του κράτος μέλος τη Μάλτα. Ε, μπορεί λοιπόν να εφαρμοστεί μια τέτοια λύση. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν. Μπορεί να, να χρησιμοποιηθεί κάτι τέτοιο στην Ισλανδία ή στην Νορβηγία. Και μην ξεχνάμε ότι σημαντικό εμπόδιο για την ε, Νορβηγία για να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ακριβώς η αλληλευτική πολιτική. Δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι προς όφελος όλων να δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε την ε, κατάσταση. Και πολύ σύντομα μια ε, ερώτηση για το ράκ της Βόρειας Θάλασσας. Από τον κύριο Άντερσον δεν άκουσα ποια είναι η θέση του για κάποια από τα βασικά ζητήματα που έχουμε μπροστά μας. Ε, αν τα τάκ και τα κότας, ε, τα τάκ ποσοστό θα πρέπει να καταργηθούν και να έχουμε ανταλλάξιμα δικαιώματα. Θα ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η θέση σας. Ε, ασχολείστε με το θέμα αυτό. Κλείνω τον κατάλογο των ομιλητών γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. <clears throat> Κρόμπατσικ, Γκούλτ, Αντρεσπαρέα, Πατρονέβες και εγώ αν έχω χρόνο θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Λοιπόν, τέρμα του καταλόγου. Κύριε Γκλόμπατσικ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε πολλές ε, απόψεις εδώ από τους ε, προσκεκλημένους μας, πολλές από τις οποίες κινούνται υπέρ μιας ε, περιφερικοποιημένης κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Κάτι επίσης το οποίο είναι σημαντικό, ίσως πιο πολύ και από την περιφερικοποίηση, ήταν το θέμα της αναγκαιότητας να αντιμετωπίσουμε τα σωστά τα αποθέματα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το να υπάρχουν περισσότερες επιστημονικές έρευνες σε σχέση με τα αποθέματα. Αν δεν έχουμε πραγματικά στοιχεία τα οποία να είναι αξιόπιστα, δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε την πολιτική μας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε τη δυνατότητα αυτή να έχουμε στερεές βάσεις και όχι να παραμείνουμε στα πλαίσια πολιτικής όπως αυτή που ισχύσε μέχρι σήμερα. Θέλω να θέσω τώρα ένα ερώτημα στον κύριο Γιώχανσεν από το Βαλτικό ΡΑΚ, γιατί μίλησε αυτό στην παρέμβασή του για την ανάγκη μιας αλλαγής στην πολιτική μας, δηλαδή να εξέλθουμε από την κυριαρχία των λόμπι. Δεν κατάλαβα τι ακριβώς τόνισε σε σχέση με τα λόμπι, αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που θέλω να θέσω και δεύτερον θέλω να ξέρω ποια είναι η δική του αξιολόγηση από την πλευρά του ΡΑΚ της Βαλτικής σε ό,τι αφορά στην βιομηχανική αλία, δηλαδή όχι αυτές που γίνονται όχι για την κατανάλωση την ανθρώπινη αλλά για βιομηχανικούς σκοπούς και ποια είναι η επίπτωση που μπορεί να έχει στα αλίευματα. Η κυτρία Πατράου Νέβες στο τέλος. Ε, ο κύριος Κούν. Κυρία Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους παριστάμενους στη σημερινή ακρόαση για τη συμβολή τους στη συζήτηση και από επαγγελματική και από επιστημονική άποψη και ιδίως την εμπειρία που μας έχουν μεταλαμβαδεύσει από την πλευρά των Περιφερειακών Συμβουλίων των ΡΑΚ. Και όλα αυτά εξυπηρετούν τον κοινό στόχο, όχι μονάχα να εξασφαλίσουμε την ύπαρξη μιας βιομάσας η οποία θα μπορεί να αλλιεύεται και στο μέλλον, αλλά να έχουμε μια πλήρη εικόνα και από τους επιστήμονες και από αυτούς που ασκούν στην πράξη την αλία. Αυτό ήταν και ο στόχος και ο λόγος δημιουργίας των ίδιων των ΡΑΚ. Είναι κρίμα ότι ο κύριος Γιώχανσεν δεν μπορούσε να μας δώσει πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τη Βαλτική. Και υπάρχει αυτή η εκδήλωση η οποία θα λάβει χώρα στην Γδίνια στις επόμενες εβδομάδες. Θα ήθελα όμως αυτό να εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία της ΙΤΣΙΣ με, την, ε, τα ΡΑΚ. Γιατί όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν κάποτε συγκεκριμένα. Υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι κινούνται προς μια κατεύθυνση, λένε ότι απειλούνται τα ψάρια μιας συγκεκριμένης περιοχής και θα πρέπει να απαγορευτούν οι αληφτικές δραστηριότητε και μετά από δύο χρόνια κάποιος έρχεται και λέει όχι έχουμε διαφορετικές απόψεις τώρα και θα πρέπει να επιτρέπεται η αλία. Είναι απαραίτητο να έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα όλοι οι οι επιστήμονες μια συγκεκριμένη θέση, να μπορούν οι επιστήμονες να βρίσκονται στα αλλιευτικά σκάφη, να βγαίνουν στην ανοιχτή θάλασσα, να βλέπουν πώς γίνεται η αλία και να μπορέσουν να ελέγξουν έτσι τις ε, μελέτες τις οποίες έχουν κάνει αυτοί πολλές φορές σε θεωρητικό επίπεδο. Αυτό ήθελα να πω. Κύριε Άντρες Μπαρέα, λοιπόν, παρακαλώ ένα ερώτημα γιατί αλλιώς θα μείνουμε χωρίς χρόνο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε ότι πάντα είμαι σύντομη. Νομίζω ότι έχει γίνει σημαντικό, έχει γίνει σαφές τώρα κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πρέπει να έχουμε τις, ε, τα επιστημονικά κριτήρια σαν κριτήριο για την πολιτική μας. Είναι απαραίτητο να έχουμε την αποκέντρωση, είναι απαραίτητο να έχουμε καλύτερα επαγγελματικά προσόντα και για τους αλείς. Είναι γεγονό πάντω ότι η γενική διαπίστωση είναι ότι η τωρινή πολιτική που βασίζεται στα συνολικά αλλιεύματα και στι ποσοστώσει δεν λειτουργεί. Και θα ήθελα να ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε μια μελέτη πιο πολύ σε βάθος για το θέμα της αλλιευτικής προσπάθειας για να προχωρήσουμε περισσότερο στον τομέα αυτό. Κύριε Πατράου Νέου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένε από τις πτυχές που τονίστηκαν εδώ από σχεδόν όλους τους παρόντες. Τα κοινά στοιχεία λοιπόν της συνένεση που υπάρχει μεταξύ μας και νομίζω ότι υπάρχει καταρχήν συμπερίληψη όλων αυτών των πτυχών στην Πράσινη Βίβλο. Λόγω ελλείψεως ε, χρόνου θα περιοριστώ σε μία προστοκία που θέλω να εκφράσω και από τη δική μου πλευρά σε σχέση με ορισμένες περιοχές, ορισμένα πελάγη και θάλασσες όπου τίθενται τόσο συγκεκριμένα ζητήματα που θα ήταν χρήσιμο να μπορούσαν να έχουν παρουσιαστεί με πιο συγκεκριμένο τρόπο για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη επαρκώς όλα αυτά τα στοιχεία. Δύο πτυχές λοιπόν θέλω να καταγράψω που ήταν θέματα αποκλίνουσών απόψεων μεταξύ των παρόντων. Το θέμα του περιορισμού στα 12 μίλια των ναυτικά μίλια των βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και εδώ δεν φαίνεται να υπήρξε συνένεση και επίσης για τα διάφορα υποδείγματα διαχείρισης μεταφερόμενα δικαιώματα αλληλείας, τάκ και ποσοστώσεις ή αλληλευτική προσπάθεια. Θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε για τα θέματα αυτά την Κομισιόν και τα ίδια τα ΡΑΚ που φυσικά δεν συμφωνούν μεταξύ τους για να γνωρίσουμε τα επιχειρήματα υπέρ και κατά σε κάθε από αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ και εγώ να θέσω δύο ερωτήματα. Ένα για τον κύριο Γκαράτ σε σχέση με το μέγιστο βιώσιμο επίπεδο απόδοσης στο οποίο εσείς αναφερθήκατε. Εσείς θεωρήσατε ότι πρέπει αυτό να εφαρμόζεται σε επίπεδο αλληλευτικής περιοχής και όχι κατά θαλάσσιο είδος. Επειδή υπάρχουν οι πολύ ιδιαίτερες λεγόμενες περιοχές όπου υπάρχουν πολλά είδη που αλλιεύονται, είπατε ότι θα είχε πιο πολύ νόημα να γίνεται έτσι. Επίσης, σε ό,τι αφορά την παράκτη αλλήλεια. Κάτι το οποίο έχει γίνει σαφέ και εδώ θέλω να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Μπαντιόλα. Ότι πρέπει να υπάρξει μια διάκριση μεταξύ τη αλληλεία ανοιχτή θάλασσα και τη παράκτεια αλληλεία. Είπατε ότι πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποιημένη αντιμετώπιση και ή δυνατόν περιφερικοποιημένη. Το ερώτημά μου είναι, εσεί πιστεύετε, κάτι το οποίο δεν το πιστεύει η Κομισιόν, ότι είναι δυνατόν να αναδιατυπωθεί, να ανακαθοριστεί η παράκτια αλληλεία, να βρούμε ένα νέο τρόπο να ε, ορίσουμε την παράκτη αλία με τρόπο ο οποίο είναι περιφερικοποιημένος και ο οποίος δεν οδηγεί σε διακρίσεις και μπορεί να ελέγχεται από τα ΡΑΚ. Και φυσικά αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τα 12 μίλια ή και παραπάνω. Το ερώτημα είναι αν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Κομισιόν και αυτούς τους οποίους απευθύνθηκαν άμεσα ερωτήσεις η Κομισιόν. Πριν απαντήσω θέλω να κάνω μια διευκρίνηση. Η Κομισιόν πιστεύει πράγματι ότι μπορεί να προκύψει ένας ορισμός της παράκτειας αλίας που να είναι προσαρμοσμένος στις συνθήκες κάθε περιοχής επί τη βάση ομοιόμορφων και κοινών κριτηρίων τεχνικού χαρακτήρα αλλά και με μια απαραίτητη ευκαμψία για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη την ανάγκη περιφερικοποίηση. Τα δύο ερωτήματα. Η συνδιάσκεψη της Κορούνια για τη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων και των επιστημόνων. Ναι, όλοι αυτοί είναι προσκεκλημένοι να συμμετάσχουν σε αυτήν την ε, συνδιάσκεψη που συνδιοργανώνεται από την Ισπανική Προεδρία και την Κομισιόν. Επίση, για το θέμα τη περιφερικοποίηση και το ερώτημα του κ. Βαλέσσα. Η περιφερικοποίηση, από την άποψη τη Κομισιόν, ε, και το είπε ο αρμόδιο επίτροπο στο Συμβούλιο των Υπουργών, την προηγούμενη εβδομάδα θεωρούμε ότι πρέπει να φτάσουμε στο απότερο σημείο που μας επιτρέπει η συνθήκη. Το πρόβλημα της ε, συνθήκης είναι ότι οι μηχανισμοί απόφασης δεν μπορούν να περιφερικοποιηθούν τελείως. Επόμενο είναι ένα θέμα αποκέντρωσης μέσα στα κράτη-μέλη και επίσης αποκέντρωση ορισμένων διαχειριστικών ικανοτήτων και δημιουργία εθνικών οργάνων που είναι παράλληλα ή παρόμοια με αυτά που έχουν δημιουργηθεί κύριε Βαλέσσα στην Βαλτική να υπάρχουν φόρουμ όπου μπορούν και τα ΡΑΚ και οι εμπλεκόμενοι και τα κράτη-μέλη όλοι οι εμπλεκόμενοι στη λήψη απόφασεων να είναι παρόντε για να συζητούνται προτάσει και να λαμβάνονται ενδεχομένω και αποφάσει όταν το επιτρέπει η συνθήκη. Αυτά λοιπόν. Η Κομισιόν υποστηρίζει την μεγαλύτερη δυνατή αποκέντρωση. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο σε αυτού οι οποίοι έχουν να αντιμετωπίσουν ερωτήσεις. Ο κ. Μπανάρ, πρώτα. Ένα, ένα λεπτό αν μπορείτε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το έγγραφο της Κομισιόν όταν αναφέρεται στο μέγιστο δυνατό εισόδημα με στη δυνατή απόδοση αναφέρεται ήδη στο σημείο αυτό και λέει ότι υπάρχει μια δυνατότητα ευρεία ερμηνεία σε ό,τι αφορά το μέγιστο βιώσιμο εισόδημα. Αυτό είναι πιο δύσκολο βέβαια στις μικτές αλίες, Γιατί όταν έχουμε διαφορετικά είδη αλλιευμάτων που αλληλεπιδρούν, είναι το, το επίπεδο αλληλεία και η ελευτική προσπάθεια δεν ανταποκρίνονται στο μέγιστο βιώσιμο επίπεδο εκμετάλλευσης κάθε συγκεκριμένου είδους. Αυτό είναι ιδιαίτερο πρόβλημα στις αλίες οι οποίες είναι πολυειδικού χαρακτήρα, περιλαμβάνουν δηλαδή πολλά ψάρια, πολλά ψαριών. Όλα αυτά λοιπόν μπορούμε να τα καταδείξουμε από επιστημονικές ε, έρευνες και θα πρέπει επομένως να έχουμε υπόψη την αρχή της προφύλαξης και να αντιμετωπίσουμε και τα κοινωνικά οικονομικά προβλήματα των αλλιέων σε αυτές τις πολιτικές περιοχές. Δίνω το λόγο τώρα στον εκπρόσωπο του ΡΑΚ της Βόρειας Θάλασσας, τον κύριο Άντερσεν. Προσπάθησα να είμαι όσο γίνεται πιο συγκεκριμένο όσον αφορά το μοντέλο αποκέντρωση. Συμφωνώ με την πρόταση της Κομισιόν, αλλά θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία και εντός του ΡΑΚ μας. Ε, και συμφωνώ με πολλούς από τους προαλήσαντες ότι δεν είναι πολύ απλό. Σίγουρα όμως, από το τελευταίο διάστημα φάνηκε ότι λόγω της ανάγκης για μικροδιαχείριση στην Κομισιόν ε, έχουν χάσει το ενδιαφέρον και πολλοί επαγγελματίες και πολλοί ε, άλλοι ενδιαφερόμενοι. Έχουμε δει ε, στατιστικές αλλά πολλοί κόσμοι έχει χάσει το ενδιαφέρον του για την πρόταση της Κομισιόν. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο με πολύ καλό τρόπο στην ε, Βόρεια Θάλασσα, στη Βαλτική. Και στην Πολωνία να πω ότι όταν τώρα μπούμε στο, ε, στην επόμενη περίοδο, επειδή γνωρίζω τη Βαλτική και την Πολωνία πολύ καλά, ξέρω ότι η Πολωνία έχει βιώσιμη αλληλεία και ε, πολύ καλό στόλο. Και στην Πολωνία συζητιέται μεταξύ αλλιέων πώς θα συνεχίσει πώς θα συνεχιστεί η εργασία αυτή. Και η και η Πολωνία ε, προτείνει πράγματα στα πλαίσια του ΡΑΚ. Εγώ πάντα ακούω τι λέει η Πολωνία και άλλα κράτη-μέλη. Μόλις όμως ε, αρχίσει να συζητιέται και η βιωσιμότητα τη αλίας θα αλλάξει πολύ η συζήτηση. Ένα λεπτό κύριε Μπαντιόλα, γιατί κάποτε πρέπει να τελειώσει και η βάρδια των διερμηνέων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Το ενοιολογικό υπόδειγμα της βιοτεχνικής αλίας το οποίο παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα. Είναι απαραίτητο να το τροποποιήσουμε και απαντώ στην κυρία Πατράου Νέβες στο ρακ του Νότου αυτό το οποίο θέλουμε είναι όχι στην αποκλειστικότητα της ε, βιοτεχνικής αλίας μέσα στα πρώτα 12 μίλια αλλά προεξάρχοντα ρόλο στη βιοτεχνική αλία χωρίς να υπάρχει πράγματι αποκλειστικότητα. Θα μας είναι πολύ σαφές. Είναι η ελευθερία πρόσβαση που είναι μια από τις βασικές ε, προδιαγραφές των συνδικών. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Εγώ πρέπει να εξασφαλίσω ότι παραμένουμε μέσα στο χρόνο που χρειάζεται. Δεν είναι πάντα εύκολο, δεν είναι πάντα ευχάριστο να εξασφαλίσω ότι όλοι πρέπει να μπορέσουν να μιλήσουν. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και θα συνεχίσουμε και το απόγευμα. Θέλω να ευχαριστήσω τους διερμηνείς για τη συνεργασία τους που είναι απαραίτητη και διακόπτω τη συνεδρίαση και πάλι στις 3 θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ σε όλους.